Colleghi, possiamo Να καθίσουμε λοιπόν παρακαλώ συνάδελφοι για να ξεκινήσουμε τις εργασίες της Επιτροπής μας. Ολοκληρώσαμε την συνάντηση των συντονιστών με λίγη καθυστέρηση για την οποία ζητώ συγγνώμη. Στην συνεδρίαση λοιπόν των συντονιστών οι συντονιστές σημερίστηκαν ε, την πρόταση να ζητήσουμε ε, από το Προεδρείο να κάνουμε πέντε επισκέψεις οι οποίες δεν θα είναι ερευνητικές αλλά θα είναι ε, επισκέψεις μελέτης σε πέντε διαφορετικές χώρες, έτσι ώστε να έρθουμε σε επαφή με συναδέλφους αντιστοίχων επιτροπών εθνικών κοινοβουλίων και να έχουμε και ανταλλαγή απόψεων με τους εκπροσώπους, με τους βουλευτές των άλλων κοινοβουλίων, άλλων χωρών. Δεχτήκαμε λοιπόν ότι θα κάνουμε ε, κάποιες επισκέψεις στην Γαλλία, την Ιταλία, την Πολωνία και μετά η Βουλγαρία ή η Ρουμανία. Επίσης ε, εγκρίθηκε η πρόταση ε, επίσκεψής μας στις 7 Δεκεμβρίου του 2010 μιας επίσκεψης λέω στο Κοινοβούλιο της Σκοτίας μετά από ε, πρόσκληση την οποία μας απίφθινε το Σκοτικό Κοινοβούλιο ε, με το σκεπτικό ότι στο Κοινοβούλιο αυτό έχουν αναπτύξει μια ιστοσελίδα εξαιρετική και επομένως θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν με τεχνογνωσία έτσι ώστε να μπορέσουμε και εμείς να δημιουργήσουμε μια αντίστοιχη ε, ιστοσελίδα. Εκείνοι έχουν χρησιμοποιήσει πολύ προχωρημένες μεθόδους και θα μπορούσαμε ενδεχομένω να έχουμε κάποια μεταφορά τεχνογνωσίας. Επίσης, αποφασίσαμε στους συντονιστές να ε, δώσουμε συνέχεια στην αναφορά του κυρίου Κλάιν για την ΑΤΜΕΔ αναφορά ε, την οποία συζητήσαμε στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Επίσης να υποβάλλουμε προφορική ε, ερώτηση κατά την έννοια αυτή προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγκρίναμε την ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασής μας με κάποιες τροποποιήσεις οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες τις εξής. Πρώτον, ψηφοφορία επί της εκθέσεως Παλιαδέλη, γιατί λόγω φυσικού λάθους χθες ψηφίσαμε επί ενός εγγράφου παλαιότερου και όχι επί της τελευταίας εκδοχής της εκθέσεως της κυρίας Παλιαδέλη. Επίσης, βάλαμε ε, στην ημερήσια διάταξη την ε, ε, έκθεση ΕΚΕΣ, της συναδέλφου ΕΚΕΣ, έτσι ώστε την επόμενη φορά να έχουμε την ανταλλαγή απόψεων, την οποία δυστυχώς δεν προλάβαμε λόγω ελήψεως χρόνου να κάνουμε χθες. Δεν έχω άλλες ανακοινώσεις σχετικές με τους συντονιστές. Μπορούμε λοιπόν να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διατάξεως. αλλά βλέπω ότι λείπει η συνάδελφος Μέρκες. Οι άλλοι συνάδελφοι... Ε, υπάρχει μάλλον κάποιος συνάδελφος που μπορεί, να μπορεί να την αντικαταστήσει, να μπορεί να παρέμβει εξ ονοματός της. Λοιπόν, από τη στιγμή που η κυρία Wallis είναι εδώ, ε, μας προτείνει ο συνάδελφος Ιτουργάης να κάνουμε μία ανατροπή λίγο της σημερινής διάταξης. Από τη στιγμή που οι συνάδελφοι Wallis και Χέφνερ είναι εδώ, μπορούμε να ξεκινήσουμε με αυτούς. Ωραία λοιπόν, θα δώσω τον λόγο ε, στην συνάδελφο Χέφνερ. Ε, ε, λοιπόν, να δώσω το λόγο στον ε, συνάδελφο ο οποίος ασχολείται με το σημείο 18. Συζητήσαμε με τον Επίτροπο Σεκοβιτς για την πρωτοβουλία των πολιτών και σήμερα απλώς θα δώσουμε μια τελική σύνθεση της χθεσινής συζήτησης. Yes, thank you. Mr. Mazzoni? No? Sorry, if it's, if it's down on the agenda... Με συγχωρείτε. Εάν είναι το θέμα προς συζήτηση στην ημερήσια διάταξη, χρειαζόμαστε λιγότερο από μία περίληψη. Θέματα που είναι στην ημερήσια διάταξη για σήμερα πρέπει να εξεταστούν σήμερα. Stiamo trattando il punto perché infatti è sulla ναι, ναι, ναι. Απλώς είπα ότι χτες συζητήσαμε το θέμα αυτό και παρουσία του Επιτρόπου. Θα κάνουμε μία σύνθεση των όσων συνέβησαν και όσων συζητήθηκαν χτες και θα κάνουμε και την κανονική συζήτηση. Yes, so, it is on the agenda today. Ναι, είναι η προσυζήτηση στην ημερήσια διάταξη σήμερα για τους δύο εισηγητές, ε, την κυρία Ούλης και εμένα, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε αυτή την συζήτηση και να ακούσουμε τις απόψεις των συναδέλφων, γιατί τώρα προχωράμε πολύ γρήγορα με την έκθεση αυτή και θέλουμε να έχουμε τις δικές σας απόψεις και τις δικές σας αντιδράσεις. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να σας ενημερώσω για κάποια ουσιαστικά θέματα και η Ταϊάννα Ουόλης μετά θα ευευθύνει το θέμα και ε, μετά αναμένουμε πολύ ε, έντονη συζήτηση. Καταρχήν, ξέρετε ότι έχουμε τώρα τέσσερις ηγητές. Δύο της Επιτροπής ε, Αναφορών και δύο της Επιτροπής ΑΦΚΟ. Γκουρμά και Λαμασούρ. Έχουμε εκπροσώπηση τεσσάρων πολιτικών κομμάτων οι περάσινοι οι το ΕΠ και οι σοσιαλιστές και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά όλοι μαζί μας. Λοιπόν, εξετάζουμε μία έκθεση παρόλο που ξέρουμε βέβαια ότι νομικά χρειαζόμαστε δύο εκθέσεις, μία για την ΑΚΤΟ, μία για την ΠΕΤΗ. Αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε είναι αυτές οι δύο εκθέσεις να έχουν το ίδιο περιεχόμενο. Για να μπορέσει λοιπόν το Κοινοβούλιο να μιλήσει με μία φωνή και να μην χρονοτριβούμε στο τέλος συζητώντα τις διαφορές μεταξύ των ε, εκθέσεων. Και γι' αυτό πάντα ε, συνεργαζόμαστε και οι τέσσερις και βρίσκουμε καλές λύσεις στα περισσότερα θέματα. Λοιπόν, θέλουμε να σας ενημερώσουμε τώρα όσον αφορά την διαδικασία καταρχήν θέλω να σας παρουσιάσω το χρονοδιάγραμμα το οποίο έχουμε κατά νου γιατί ο στόχος μας είναι να είμαστε έτοιμοι με την ε, νομοθεσία αυτή για τα τέλη του έτους. Ένας από τους λόγους είναι ότι αυτή είναι μία από τις έντονες υποσχέσεις που δίνονται από τις συνθήκε Λισαβόνας και δεν έχουν ακόμα υιοθετηθεί. Μετά θα έχουμε μια συνάντηση με την Προεδρία μέχρι τα τέλη του έτους και θα πρέπει να ξεκινήσουμε πολλές συζητήσεις μαζί σας. Όταν περάσουμε και στη νέα Προεδρία, στην Ουγγρική, δηλαδή, Και γι' αυτό εμείς από δική μας κοπιά, από πλευρά Κοινοβουλίου, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην αποδυναμώσουμε, να μην χρονοτροβήσουμε, να προχωρήσουμε στο γρηγορότερο δυνατόν. Η πρόταση μας είναι στις 9 Νοεμβρίου, εδώ στην Επιτροπή ε, Αναφορών, να παρουσιάσουμε ήδη ένα σχέδιο έκθεσης. μπορεί να συζητήσει και να ψηφίσει η Επιτροπή Αναφορών και ταυτόχρονα να δοθεί στους ε, εισηγητές μία εντολή για διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και με την Επιτροπή, την Εκταλιστική Επιτροπή. Αυτό προσπαθούμε λοιπόν να πετύχουμε είναι να συμβεστούμε όσο δεν τον γίνεται πριν υποβληθεί το σχέδιο της ε, ε, έκθεσης στο τέλος στο Κοινοβούλιο και να έχουμε μία πρώτη συμφωνία για την πρώτη ανάγνωση τη, σχετικά με την, ε, με την υπόθεση αυτή. Και κατόπιν θα έχουμε επαφέ με την Κομισιόν και με το Συμβούλιο και ανάλογα με τα αποτελέσματα μπορούμε να σας το υποβάλουμε ξανά στην Επιτροπή εδώ αναφορών και να ψηφίσουμε στις 22 Νοεμβρίου Και αν χρειάζεται και άλλη μία συνεδρίαση για να ψηφίσουμε, θα προβλέπουμε στις 13 Δεκεμβρίου και η τελική ψηφοφορία στην Αλαμέλεια για την πρωτοβουλία των Ευρωπαίων πολιτών να γίνει στις 16 Δεκεμβρίου. Και έτσι θα ολοκληρώσουμε πριν από τα τέλη του έτους. Τώρα γενικά όσον αφορά την ε, γενική προσέγγιση των τεσσάρων συγητών. Η προσέγγιση προβλέπει να πάρουμε την πρόταση της Κομισιόν και να προσπαθήσουμε να το καταστήσουμε πιο εύχρηστη για τους πολίτες και πιο αποτελεσματική. Γιατί πολλά προβλέπονται αυτό το σχέδιο του κανονισμού που δεν είναι πολύ πρακτικά εφαρμόσιμα, δεν είναι φιλικά προς τον χρήστη και θα οδηγήσει σε πολύ δυσαρέσκεια θα πρέπει να μπορέσουμε να καλέξουμε τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν αυτό το νέο μέσο, την πρωτοβουλία δηλαδή των Ευρωπαίων πολιτών, για να μπορέσουν να διατυπώσουν τις δικές τους επιθυμίες προς την Κομισιόν, προς το Κοινοβούλιο. Δεν θα πρέπει λοιπόν να τους να καταστήσουμε τη ζωή τους δύσκολη, να έχουμε μεγαλύτερη γραφειοκρατία, αλλά ένα σύστημα και ένα μέσο ε, το οποίο να είναι εύκολα προσιτό. Εδώ λέγεται. Θα πρέπει οι πολίτες να συλλέξουν 300.000 υπογραφές, να σταματήσουν να συλλέγουν, ε, να εξετάσει η Επιτροπή κατά πόσον αυτό είναι ε, αποδεκτό ή όχι και εάν ναι να συνεχίσουν, εάν όχι να σταματήσουν. Δεν είναι λογικό να ξεκινήσει η διαδικασία και όταν έχουν μαζέψει τι 300.000 υπογραφές να τους πούνε ναι μπορείτε ή δεν μπορείτε. Όχι, αυτό θα πρέπει να γίνεται στην αρχή. Και ο κανονισμός εδώ θα πρέπει να είναι πιο απλός, πιο ακριβής. Η Κομισιό θα εξετάζει κατά πόσο είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αρμοδιότητα της ε, ε, Κομισιό να υποβάλει ε, μια τέτοια πρόταση κατά πόσο δεν είναι αντίθετο με τις ε, βασικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αν όλα αυτά τηρούνται, τότε θα μπορούν να αρχίσουν τη δικασία ε, υπογραφών. Και το αποδεκτό θα γίνει άμα μαζέψουν τουλάχιστον ένα εκατομμύριο υπογραφές. Αυτά για τις γενικές γραμμές και το χρονοδιάγραμμα και η κυρία Βόλης τώρα θα συνεχίσει και θα σας παρουσιάσει τις, απο... τις ε, απόψεις μας και μετά μας ανοιχτεί στις δικές σας παρατηρήσεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Βόλης. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έφνερ πολύ καλά παρουσίασε την κατάσταση που βρισκόμαστε. Συνεργαζόμαστε με τέσσερις εισηγητές από τέσσερις διαφορετικές κοινοβουλευτικές επιτροπές και ομάδες. Πάνε καλά τα πράγματα. Πάντως, όσο προχωράμε, βλέπουμε ότι διάφορες λεπτομέρειες πρέπει να λυθούν και εκεί προσπαθούμε να βρούμε λύσεις που να είναι αποδεκτές από όλους, που να νιώθουν όλοι καλά με αυτές. Έχουμε τη φιλοδοξία και πρέπει να την έχουμε να τελειώσει αυτή η διαδικασία μέχρι τα τέλη της χρονιάς για όλους τους λόγους που ακούσαμε και πριν. Δεν θα πρέπει να γίνει όπως έχει ξαναγίνει, δηλαδή να παραβλεφθούν τα δικαιώματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όχι, πρέπει να φροντίσουμε να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο μας για να ακουστεί η φωνή μας και να έχουμε μια πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών φιλική προς τους Ευρωπαίους πολίτες. Έχουμε λοιπόν τη φιλοδοξία και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Αν όμως υπάρχουν δύσκολα ζητήματα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να κρατήσουμε σκληρή στάση απέναντι στα άλλα θεσμικά όργανα. Είπαμε ότι η προσέγγιση μας είναι να βρούμε μια φιλική για τον Ευρωπαίο πολίτη προσέγγιση. Και αυτό το επιχείρημα κερδίζει έδαφος, πρέπει να ξέρετε, και στις άλλες πλευρές. Ιδιαίτερα για το πρώτο βήμα καταχώρησης της πρωτοβουλίας. Αντί να πρέπει να συλλέγονται πρώτα πάρα πολλές υπογραφές, εμείς πιστεύουμε ότι τέσσερις άνθρωποι από... Συγγνώμη, 7 άνθρωποι από 7 διαφορετικές χώρες μέλη φτάνουν για να έχουμε ε, το ξεκίνημα της διαδικασίας. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει εγγύηση ότι πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό θέμα, ότι είναι κάτι που συζητιέται στην Ευρώπη και βάσει αυτού να ξεκινάμε. Μετά η Επιτροπή να το κοιτάζει. Όσοι ήταν εδώ χτες θα ακούσανε τη χτεσινή συζήτηση με τον Επίτροπο, ο οποίος τόνισε το θέμα της, του διοικητικού ελέγχου. Ο έλεγχος που θα γίνεται θα είναι διοικητικό, για να μην μπαίνει σε δύσκολη θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να είναι και κριτής και κρινόμενος. Ακούστηκαν διάφορες ενδιαφέρουσες ιδέες χτες, να έχουμε μια επιτροπή σοφών ή κάποιον άλλον που θα κρίνει στην αρχή. Κατά τη γνώμη μας αυτό περιπλέκει την όλη διαδικασία χωρίς λόγο. Θέλουμε να είναι μια απλή και ξεκαθαρή διαδικασία. Αυτό είναι το όλο ζήτημα. Το ακούσατε και πριν. Θέλουμε να είναι μια ανοιχτή προσφορά στους Ευρωπαίους πολίτες, ώστε να μπορούν εύκολα να ασχολούνται με την πολιτική ζωή της Ευρώπης οι πολίτες μας. Συγχρόνως όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι μια σοβαρή δυνατότητα για να μπορέσουμε καλύτερα να ετοιμάσουμε την ατζέντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μέλλον. Αυτό είναι. Και από μόνο του είναι πολύ σημαντικό. Αλλά είναι αυτό, δεν είναι τίποτα παραπάνω. Μην το κάνουμε λοιπόν πιο περίπλοκο από ό,τι χρειάζεται. Επαναλαμβάνω και τα δύο πράγματα που είπα χτες από αυτού. Πιστεύουμε και οι τέσσερις εισηγητές συμφωνούμε ότι θέλουμε να μπορούμε να συμπεριλάβουμε οποιοδήποτε πολίτη πάνω από τα 16, 16 ετών. Γιατί οποιοδήποτε από τα 16 και πάνω πρέπει να έχει το δικαίωμα να υπογράφει μια πρωτοβουλία. Γιατί αυτό κάνουν. Δεν κάνουν τίποτα άλλο. Υπογράφουν την πρωτοβουλία. Είναι σημαντικό γιατί έτσι οι νέοι προετοιμάζονται καλύτερα να κάνουν το μεγαλύτερο βήμα που είναι να φτάσουν στην ηλικία ε, κατά την οποία μπορούν και να ψηφίσουν. Πρέπει να είμαστε ανοιχτοί λοιπόν. Και εμείς στην Επιτροπή μας μπορούμε να αναρωτηθούμε μήπως θα θέλαμε η διαδικασία αυτή να είναι ανοιχτή για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες οποιασδήποτε ηλικία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μεταξύ μας οι διάφοροι ευρωβουλευτές συμφωνήσαμε για τα 16. Και έπειτα να υπάρχει το ίδιο όριο για όλες τις χώρες. Να μην είναι διαφορετικό το όριο στη μία χώρα και διαφορετικό στην άλλη. Αυτό ήταν το πρώτο. Το δεύτερο τώρα που θα είναι δύσκολο και επίμαχο. Αυτό είναι η ιδέα που υπάρχει σε ορισμένες χώρες για να θεωρούν έγκαιρες ε, οι αιτήσει θα πρέπει να καλύπτονται από συγκεκριμένο αριθμό υπογραφών. Θα έλεγα ότι οι συνάδελφοι καλό θα ήταν να κοιτάξουν μια έκθεση που έχει ετοιμάσει η ΚΑΣ και που δείχνει πόσο δύσκολο είναι να ζητάμε στοιχεία ταυτότητας για κάθε άτομο που θέλει να υπογράψει μια πρωτοβουλία. Στη χώρα μου, για παράδειγμα, οι άνθρωποι δεν θέλουν να τους ζητάτε τα στοιχεία ταυτότητάς τους. Και νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσει το Κοινοβούλιο και να πει ότι δεν χρειάζονται στοιχεία ταυτότητας, αριθμοί διαβατηρίων ή δεν ξέρω τι, κάθε φορά που κάποιος θέλει να υπογράψει μια πρωτοβουλία. Ας μείνει απλή αυτή η διαδικασία για να ε, φροντίσουμε έτσι να έχουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο που θα συμμετέχει σε αυτές τις πρωτοβουλίες. Αυτά. Πρέπει να είναι ξεκάθαροι κανόνες βέβαια πώς προχωράει η διαδικασία. Τι πρέπει να κάνει κανείς για να ξεκινήσει μια πρωτοβουλία. Πρώτα απ' όλα, εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μπορεί ξεκάθαρα να απαντήσει σε αυτά με τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου. Πάντως θέλουμε η Επιτροπή να είναι υποχρεωμένη να απαντάει στην ίδια προθεσμία και με τον ίδιο τρόπο όπως απαντάει και σε ένα νομοθετικό ψήφισμα, μια νομοθετική πρωτοβουλία. Πρέπει να ανταποκρίνεται δηλαδή στις προτάσεις αυτές πρωτοβουλίας πρέπει να ισχύουν οι ίδιοι κανόνε κανόνες δηλαδή για τις πρωτοβουλίε των πολιτών όπως ισχύουν και εδώ. Η Επιτροπή μας τώρα πρέπει να δει εμείς πώς θα συμμετέχουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν χρειάζεται να συμμετέχουμε στους ε, κανονισμούς και στους κανόνες που θα ισχύουν, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα συμμετέχουμε και να υπάρχει περιθώριο για την δικιά μας την εμπλοκή στην διαδικασία αυτή στο μέλλον. Ευχαριστώ. Το λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τους δύο εισηγητές μας. πολύ ενδιαφέροντα τα σημεία τους. Μέχρι τώρα βρήκα και τους δύο συγγητές ανοιχτούς, πρόθυμους να μας ακούσουν. ιδέα όμως για τη συμφωνία πρώτης ανάγνωσης και το χρονοδιάγραμμα με ενοχλεί πολύ. Τότε εξακολουθούν να γίνονται συζητήσεις και ότι τελικά είναι οι συγητές και η Επιτροπή οι συγητές και άντε πάλι συγητές και δεν υπάρχει feedback από πιο έξω, δεν μ' αρέσει. Αν λέει η μερίσια διάταξη συζήτηση της πρότασης, σημαίνει συζήτηση της πρότασης. Δεν σημαίνει έχουμε ένα σχέδιο και το ψηφίζουμε. Συγχρόνως. Εμένα με πιέζει αυτό. Κοιτάξτε, εγώ συμμετείχα για μια νομοθετική διάταξη ως εισηγήτρια. Είχαμε πολύ στενή προθεσμία, ήταν νομοθετική πράξη και έπρεπε οπωσδήποτε να το κάνουμε. Εντάξει. Δεν λέω ότι με κατά των συμφωνιών πρώτης ανάγνωσης, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες που δεν έχουν ιδέα. Τώρα ξεκινάνε με αυτό. Και νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Λέτε ότι αυτό είναι ένα από τα πράγματα στη συνθήκη της Λισαβόνας που δεν έχει αρχίσει ακόμα να εφαρμόζεται. Ναι, αλλά είναι ένα κάτι. Είναι όμως κάτι που ακριβώς πρέπει να δείξει ότι οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν. Ε, οπότε εδώ ούτε οι πολίτες μπορούν να συμμετέχουν, ούτε οι σκιώδεις εισηγητές δεν μπορούν να συμμετέχουν. Αν δεν έχουν έγκαιρα μπροστά τους το τι συζητιέται, το ποιες είναι οι προτάσεις που συζητιούνται κλπ. Πόσο μάλλον να υπάρχει στην ημερήσια διάταξη και να μας λέτε «Μα το συζητήσαμε χτε. Οπότε αφού το συζητήσαμε χτε, δεν χρειάζεται να το ξανασυζητήσουμε σήμερα. Θα ήθελα πιο συχνές συναντήσεις και επαφές με τους ε, εισηγητές και να υπάρχει feedback από τις διάφορες ε, συνεδριάσεις που γίνονται, να μπορούμε να συζητάμε τη διατύπωση. Ε, τίποτα από όλα αυτά δεν γίνεται όμως. Και εγώ θα περίμενα στο μέλλον ότι θα γινόταν, αλλά με το χρονοδιάγραμμα αυτό αποκλείεται. Οπότε ούτε οι πολίτε θα συμμετέχουν, ούτε εγώ δεν θα μπορώ να συμμετέχω που είμαι σκιώδη εισηγήτρια. Δεν είναι ρεαλιστικό. Έβαλα το όνομά μου πρόσθετα, αλλά τελικά αυτό μόνο θα είναι, ένα όνομα. Συζητήσεις που να μπορεί να έρθει ο κόσμος και να μας πει ναι, βλέπουμε τι συζητιέται, ποια είναι η διατύπωση. Εμεί πιστεύουμε ότι αυτή η πρόταση πρέπει να γίνει η άλλη, αυτή η τροποποίηση. Δεν γίνεται. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, μου αρέσει η προσέγγιση των εισηγητών όσον αφορά το περιεχόμενο. Κάποια πράγματα που εγώ θα πρόσθετα και που έχουν συζητηθεί αλλού, σε άλλες επιτροπές, είναι ότι θέλουμε οι πολίτες να έρθουν πιο κοντά στην Ευρώπη. Πολίτες σημαίνει πολίτες αυτοί που μπορούν να ψηφίζουν και όχι οι υπόλοιποι δηλαδή. Ναι, αλλά όταν λέμε θέλουμε να είμαστε πιο κοντά στους Ευρωπαίους πολίτες, εννοούμε κάθε κάτοικο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ή έτσι θα έπρεπε να εννοούμε. Και όχι μόνο αυτούς που ψηφίζουν. Εγώ δεν λέω ότι θα παίρνω το λόγο στις συνεδριάσεις που γίνονται μεταξύ των εισηγητών, αλλά τουλάχιστον να μπορώ να παρακολουθώ. Να είναι εκεί και οι σκιώδες, να είναι παρόντες, να μην τα μαθαίνουν από δεύτερο χέρι και να έχουν χρόνο και οι πολίτες να λένε τη δικιά τους ε, άποψη. Εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά γίνονται και κλεισμένων των θυρών και μακριά από τον πολίτη. Θα ήθελε η δικιά μας Επιτροπή για την πρωτοβουλία αυτή τουλάχιστον να μην ακολουθεί μια τέτοια διαδικασία. Ο κύριος Μποσινάρου, ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω δύο σύντομα σχόλια. Πρώτον, ενθαρρύνομαι μετά από αυτά που είπε χτες ο Επίτροπος και οι ξέχοντες εδώ συνάδελφοί μας που μας εξηγούν πώς έχουν τα πράγματα εν ώψη συμβιβασμού. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την έκθεσή μας. Αν υπάρχει τέτοια δέσμευση από κάθε πλευρά για συμβιβασμό, τότε θα έχουμε καρποφόρες εργασίες. Και εγώ είμαι ότι έχοντας τέσσερις μεγάλες πολιτικές ομάδες που συμμετέχουν και που ετοιμάζουν την έκθεση αυτή θα τα καταφέρουμε. Συγχρόνως έχουμε και έναν επίτροπο ο οποίος είναι δεσμευμένος υπέρ ε, μιας αποτελεσματικής πρωτοβουλίας Ευρωπαίων πολιτών. Άρα στο τέλος θα έχουμε μια πολύ πετυχημένη υπόθεση, success story, για μια τέτοια νομοθεσία. Για το χρονοδιάγραμμα τώρα και τις προθεσμίες. Ξέρω ότι είναι δύσκολα τα πράγματα πρέπει να είναι ένα πραγματικά ελβετικό ρολόι που θα δουλεύει και θα ρυθμίζει την κατάσταση. Αν θέλουμε το 2011 η πρωτοβουλία Ευρωπαίων πολιτών να είναι με σάρκα και οστά, πρέπει να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Πώς μπορούν να συμμετέχουν οι σκιώδεις και εγώ είμαι σκιώδης εισηγητής για τη δικιά μου την ομάδα. Με δύο τρόπους μπορεί να γίνει αυτό. Πρώτον, οριζόντιες ομάδες εργασίας ή κάτι αντίστοιχο στις πολιτικές μας ομάδες προκειμένου αυτές να ενημερώνονται από τους συνεισηγητές. Είναι ο μόνος τρόπος σε καθημερινή βάση να έχουμε ενημέρωση για τις διαπραγματεύσει και τις προτάσεις και έτσι μετά να προετοιμάζουμε και τις πολιτικές μας ομάδες κατάλληλα για το περιεχόμενο των προτάσεων. Δεύτερον, θα πρότεινα στην Πρόεδρο και στους αξιότιμους συν να έχουν τακτικά συναντήσεις με τους σκιώδεις εισηγητές εδώ στην Επιτροπή Αναφορών. Έτσι κανένας δεν αποκλείεται. Κανένας δεν μένει έξω από τις εξελίξεις. Και, και με αυτό θα τελειώσω, αν θα μπορέσουμε να έχουμε πολιτική στήριξη ευρεία, Σημαίνει δηλαδή πολλές ψήφους υπέρ της έκθεσης. Αυτόματα θα έχουμε και μεγαλύτερο λόγο στις διαπραγματεύσεις που θα κάνουμε με την Επιτροπή και το Συμβούλιο. Είναι ο μόνος τρόπος για να κάνουμε την πρωτοβουλία αυτή ρεαλιστική και ένα σπουδαίο εργαλείο στην διάθεση των Ευρωπαίων πολιτών. Αλλιώς θα έχουμε χάσει χρόνο. Εγώ όμως πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Και πάλι χαίρομαι για την δέσμευση που έχουν αναλάβει οι, οι μας να συνεργάζονται με τους άλλους συγητές και να μας ενημερώνουν. Να ξέρετε ότι μπορείτε να βασιστείτε στη στήριξή μας. Σας ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Γιάρη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Πρώτα απ' όλα όλοι θέλουμε αυτή την πρωτοβουλία των πολιτών, των Ευρωπαίων πολιτών. Όλοι το θέλουμε. Και θα πρέπει, όπως είπαν και άλλοι συνάδελφοι, η εργασία μας να στρέφεται και να αφορά τους Ευρωπαίους πολίτες, άνδρες και γυναίκες, έτσι ώστε και η ε, κοινή γνώμη ε, να ε, σταματήσει να μας βλέπει σαν αυτούς που σταματούν όλες τις διαδικασίες και πρέπει να είμαστε εδώ για τους πολίτες. Τώρα, το χρονοδιάγραμμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και αν θέλουμε να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα, πρέπει οπωσδήποτε οι σκιώδεις εισηγητέ να θεωρηθούν κατά κάποιο τρόπο οι σύνδεσμοι με τις πολιτικές ομάδες. Γιατί ε, αυτές τις συμβαστικέ λύσεις θα πρέπει εμείς τελικά να τις πουλήσουμε εντό εισαγωγικών, να τις περάσουμε στις πολιτικές μας ομάδες. Οι σκιώδεις εισηγήσεις είναι πολύ σημαντικές στην παρούσα περίπτωση. Και όπως είπε και ο συνάδελφος Μποστινάρο, όπως έχει πάρα πολύ δίκιο, οι εισηγητές θα πρέπει σε, τακτικές, σε, σε τακτά διαστήματα να ανταλλάσσουν απόψεις με τους κοιόδους εισηγητές, γιατί διαφορετικά δεν θα προχωρήσουμε γρήγορα και ε, τελικά να αποφασίσει, το χειρότερο δηλαδή, να αποφασίσει η Ολομέλεια ότι η έκθεση δεν είναι ακόμα όριμη. Επομένως, εγώ ε, θέλω να δεχθούμε το, την, ε, το χρονοδιάγραμμα και εγώ θα ήθελα ο σκιώδης συγητής μου να έρχεται τακτικά σε επαφή μαζί μου. Τώρα, ε, εάν θέλουμε να ορίσουμε το 16ο σαν έτος ε, όριο και αν αυτό είναι προς το καλό των πολιτών, ναι. Αλλά το ζήτημα είναι ε, να κάνουμε ό,τι γίνεται καλύτερο για τους ε, πολίτες. Δηλαδή, εάν καταλάβουν κάποια στιγμή ότι ε, στο 30-40% υπάρχουν των αιτήσεων, υπάρχουν, των αναφορών συγγνώμη, υπάρχουν προβλήματα, εάν έχουμε διπλές υπογραφές. Also bitte ich auch um den Kompromiss. Und die dritte Anmerkung, was mich immer beschäftigt ε, εάν δουν ότι υπάρχουν επικαλύψεις, διπλές υπογραφές, ε, τότε ε, θα έχουν και μία δυσκολία να μας πιστέψουν. Πιστεύω λοιπόν ότι και για τις πρωτοβουλίες υπάρχει πάντα ένα ελάχιστο όριο υπάρχουν ε, και αυτές ε, οι οποίες ε, περνούν ξιστά. Ξέρετε, σαν τον κόλ που περνάει ξιστά από το δοκάρι. Και τελικά δεν μπαίνει βέβαια. Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι οι πρωτοβουλίες οι οποίες από λίγο δεν καταφέρνουν να περάσουν να μην χαθούν τελείως. Γιατί είναι κρίμα και επαναλαμβάνω ότι θα πρέπει να υπάρχει, αυτό το σημειώνω και το υπογραμμίζω, καλή συνεργασία ανάμεσα στους ε, ε, εισηγητές, στους κοιόδης εισηγητές, γιατί αυτό που θέλουμε είναι να προχωρήσει πραγματικά αυτή η πρωτοβουλία. Τι θέλουμε όντως. Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε να απαντήσετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά αυτή τη φορά, λέει ο κύριος Αφνέρ. Θα απαντήσω πρώτα στην κυρία Ντεμπράν. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά αυτό που λέτε. Και ουσιαστικά συμφωνώ μαζί σας. Αν αυτό που προτείνουμε εδώ σαν διαδικασία σημαίνει ότι μόνο μερικοί συμμετέχουν στις διαπραγματεύσεις και οι υπόλοιποι όχι, ε, είμαι ο πρώτος που θα αντιτεθώ. Ο πρώτος. Όταν η Νταϊάννα Βόλης λοιπόν και εγώ δεχτήκαμε να αναλάβουμε ως εισηγητές, είχαν ήδη ξεκινήσει διαπραγματεύσει και είπαμε «Α, όχι, πρέπει να είναι ανοιχτά τα πράγματα, όλοι να συμμετέχουν, να μην είναι κλειστές οι διαπραγματεύσεις και όλοι και εσείς και όλοι να μπορούν να ενημερώνονται και εμείς να μπορούμε να σας μεταφέρουμε τις σκέψεις μας και εσείς να μας λέτε τις δικές σας, να τις ενσωματώνουμε στις διαπραγματεύσεις και έτσι να προχωρήσουμε. Εμείς έχουμε προσκαλέσει όλους τους σκιώδεις συζητητές από όλες τις κοινοβουλευτικές επιτροπές και τους ζητήσαμε να μας στείλουν τις ανησυχίες τους και να συνεχίσουν να το κάνουν αυτό. Η διαδικασία αυτή πρέπει να είναι μια διαδικασία ολόκληρη του Κοινοβουλίου. Εννοείται κάποιος πρέπει να είναι παρόν. Δεν μπορούν όλοι να είναι παρόν, αλλά οι προτάσεις δεν γίνονται ρήμιν σας. Αυτά λοιπόν που σας παρουσίασα σήμερα σημαίνουν τακτικές επαφέ με τους σκιώδε συζητητέ και τις πολιτικές ομάδες. Αλλιώς ούτε για μένα είναι αποδεκτή μια διαφορετική διαδικασία. Τώρα, αν δεν καταφέρουμε να πετύχουμε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση, θα πρέπει να ακολουθήσουμε τη συνήθη διαδικασία. Συμφωνία σημαίνει αυτό που σημαίνει. Συμφωνία σημαίνει ότι το Κοινοβούλιο θα πει ναι για ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Αν δεν πει ναι το Κοινοβούλιο, τότε το Κοινοβούλιο θα υιοθετήσει μια έκθεση και μετά θα κάνει διαπραγματεύσεις. Έχω την αίσθηση ότι πολλά θέματα δεν θα λυθούν παρά μόνο με συνεχείς συζητήσεις. Για παράδειγμα, μια ε, επιτροπή ζωτάει από τα κράτη-μέλη. Ποια έγγραφα χρειάζεστε εσείς για να επαληθεύετε ότι κάποιος που υπογράφει την πρωτοβουλία έχει όντως δικαίωμα να την υπογράψει. Και μερικές φορές τα κράτη-μέλη στέλνουν τεράστιο κατάλογο με αιτιολογικά, με έγγραφα. Εμείς μετά είπαμε, ναι, αλλά πώς σήμερα επαληθεύετε όταν έχετε πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο πολιτών σας, πώς επαληθεύετε τις υπογραφές. Και εκεί σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη αποδείχθηκε ότι δεν τα χρειάζονται όλα αυτά τα έγγραφα, οπότε τώρα διαπραγματευόμαστε να σκεφτούμε, «Ε, τα πραγματικά τα χρειαζόσαστε όλα αυτά τα δικαιολογητικά. Οι συζητήσει, δηλαδή είναι κάτι αναγκαίο έτσι αλλάζουν οι θέσεις, έτσι προχωράμε. Δεν πρέπει να μένουμε σε μια αποτυχία, χρειάζονται συζητήσεις για να αλλάξει η κατάσταση. Τέλη Μαρτίου έκανε η Επιτροπή την πρότασή της, αλλά συνεχίζει να σκέφτεται. Συνεχίζει να εξετάζει πώς μπορεί να βελτιωθεί η πρόταση αυτή, γιατί η πρόταση έπρεπε να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και επιδέχεται βελτιώσεις και πρέπει να βελτιωθεί. Αυτά λοιπόν που εμείς προτείνουμε εδώ τώρα περνάνε και φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή η οποία τα αντιμετωπίζει πολύ θετικά. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τις διάφορες απόψεις. Και τότε θα προχωρήσουμε. Αν δούμε όμως ότι αυτό δεν γίνεται, τότε το Κοινοβούλιο είναι ελεύθερο να πάσα στιγμή να πει όχι, δεν θέλουμε τη συμφωνία, δεν βλέπουμε να μπορεί να επιτευχθεί η συμφωνία και να επιστρέψουμε στην συνήθη διαδικασία. Σήμερα στην Ευρώπη έχουμε κυβερνήσεις που διαφέρουν πολύ μεταξύ τους και αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο. Υπάρχει λοιπόν ανησυχία μήπως έχουμε στην Ουγγαρία για παράδειγμα ε, τεράστια στροφή. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει λοιπόν αν καθυστερήσουμε και περιμένουμε πάρα πολύ και υπάρχουν ε, τεράστιες αλλαγές εκεί. Αυτό είναι άλλος ένα λόγος για τον οποίο θέλουμε γρήγορα να καταλήξουμε σε αποτελέσματα. Πέρα από το ότι το θέλουν οι πολίτες να προχωρήσουμε γρήγορα. Και κάτι τελευταίο. Όλα όσα είπατε στις διάφορες συναντήσεις που είχαμε με τους σκιώδεις εισηγητές αλλά και στις συνεδριάσεις μας εδώ, τα έχουμε συμπεριλάβει. Το θέμα ε, των ε, κατοίκων, το να είναι οι κάτοικοι, αυτή είναι η δικιά μας η θέση στις διαπραγματεύσεις πια. Αυτό που έχετε πει εσείς. Γι' αυτό σας λέω ότι είμαστε ανοιχτοί στις δικές σας τις θέσεις και τις θέλουμε, τις θέσεις σας και όλα. Ευχαριστώ. Momento, la collega ε, ε, κοιτάξτε, κυρία Γόλης, περιμένετε λίγο. Έχουν, έχουμε ένα άλλο αίτημα ε, να μιλήσει πρώτα συνάδελφος και μετά. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη αλλά θα ήθελα και να ευχαριστήσω τους εισηγητές γιατί βλέπω ότι το ζήτημα το οποίο εθιγεί όσον αφορά τη συνεργασία με τους σκιώδεις εισηγητές με βρίσκει απολύτω σύμφωνη. Συμφωνώ και με αυτά που είπε ο κ. Χαεφνέρ, δηλαδή είχαμε ένα πρόβλημα γιατί το πρώτο κείμενο ήταν προχωρημένο σε σχέση με το δικό μας κατά κάποιο τρόπο αλλά πρέπει να πω ότι οι δύο εισηγητές μας ε, μας συνάντησαν, ε, ήθελαν ανταλλαγή απόψεων μαζί μας. Ε, μία πρώτη δυσκολία λοιπόν αυτή της, του προσχεδίου ε, ξεπεράστηκε. Θα θέλαμε λοιπόν ο διάλογος να γίνει διαρκή, σταθερός και επικοδομητικός. Γιατί άλλωστε μέσω αυτού του διαλόγου καταφέραμε να προσεγγίσουμε τις θέσεις μας. Ε, ξέρετε, εγώ έκανα ε, έναν πίνακα που συγκρίνει τα δύο κείμενα. Στην αρχή βλέπαμε πάρα πολλά στοιχεία τα οποία φαίνονται να μην συνδυάζονται καθόλου. Αλλά Χάρη στην διαρκή προσπάθεια των εισηγητών, χάρη στο διάλογο, καταφέραμε να έχουμε μια κοινή θέση. Γι' αυτό λοιπόν είναι εξαιρετικά σημαντικό εμείς ως Ευρωπαίοι βουλευτές να έχουμε μια θέση τέτοια που θα αποτελέσει ισχυρό, ηχηρό μήνυμα προς τους ε, ε, πολίτες της Ευρώπης. Ε, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, βεβαίως θα συμφωνήσω, γιατί αυτή η πρωτοβουλία των πολιτών ανακοινώθηκε με πολύ θόρυβο πριν από ένα χρόνο και παραπάνω. Έχουν αρχίσει ήδη να αναρωτιούνται οι πολίτες τι γίνεται με αυτό. Λοιπόν πρέπει να αναλάβουμε τις ε, ευθύνες μας ε, να τους σεβαστούμε ε, και να σεβαστούμε και τις θέσεις μας. Όπως είπε και ο Σλάνφος Χέφνερ, η Επιτροπή ήδη εξέφρασε την άποψή της. Ακούσαμε χθε τον κύριο ε, Σεύκοβιτς, ακούσαμε ότι ορισμένα πράγματα εξακολουθεί να τα συζητάει η Επιτροπή, αλλά ε, εμείς πρέπει να υπεραμεινθούμε της δικής μας ε, θέσεως. Ε, ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους συναδέλφους, να δείξω την έμπρακτη ελληνική μου μαζί τους και να σιγουρευτούμε όλοι ότι θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε μαζί έτσι ώστε να σεβαστούμε και το χρονοδιάγραμμα αφενός και για να μπορέσουμε να έχουμε κοινή θέση αφετέρου. Η κυρία δεν θέλω να σας καθυστερήσω. Ευχαριστώ πάντως τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους και να καθισκάσω την κυρία Μπροϊν. Και εγώ μισώ την πρώτη ανάγνωση όπως και εσείς. Αλλά μερικές φορές είμαστε σε μια κατάσταση που έχουμε την φιλοδοξία να προχωρήσουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα και πρέπει να το κάνουμε με εσά και με τη στήριξή σας. Γι' αυτό λοιπόν ζητάω, δεν ξέρω αν είναι εφικτό, αν η γραμματεία μπορεί να μας βοηθήσει σε αυτό, μέσα στο χρονοδιάγραμμα που έχουμε ήδη να προβλέψουμε τη δυνατότητα συνάντησης με τους σκιώδεις εισηγητές μας, έτσι ώστε να είναι σίγουρο ότι συμμετέχετε πλήρως στη διαδικασία. Γιατί σας διαβεβαιώ δεν υπάρχει καθόλου η πρόθεση να σας αποκλείσουμε. Χρειαζόμαστε τη στήριξή σας. Χρειαζόμαστε όσο γίνεται πιο ευρεία στήριξη. Μην ξεχνάτε ότι μία συζήτηση κάναμε με τα άλλα δύο θεσμικά όργανα και χτες το ακούσατε και από τον Επίτροπο. Δεν έχουμε προχωρήσει δηλαδή πολύ χωρίς εσάς, μην νομίζετε. Και έχουμε θετικά μηνύματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι έρχεται στις θέσεις μας. Οπότε το Κοινοβούλιο με τους τέσσερις εισηγητές δείχνει να είναι αποτελεσματικό στις διαπραγματεύσεις. Τώρα θέλω να πω κάτι στον κύριο Γιάρε, ο οποίος έθεσε το θέμα των πρωτοβουλειών που τελικά δεν περνάν τον πύχη, την πάρα. Βάζουμε κανόνες για τις πρωτοβουλίες αυτές που πρέπει να είναι σαφέστατες για να έχει νόημα η διαδικασία. Συμφωνώ όμω μαζί σας για το ότι πρέπει να υπάρχει κάποια θέση αναδίπλωσης έτσι ώστε η Επιτροπή μας να μπορεί να χειριστεί τις πρωτοβουλίες που ίσως δεν περνάνε σαν πρωτοβουλίες Ευρωπαίων πολιτών και να μπορεί να κάνει κάτι με αυτές. Να βρούμε δηλαδή μια τέτοια δυνατότητα. Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους εισηγητές και τους σκιώδεις εισηγητές και όλους όσους πήραν το λόγο. Πιστεύουμε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και όλα αυτά που ακούστηκαν είναι εξαιρετικά ωφέλιμα και οπωσδήποτε θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας. Μεγαλύτερη συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στη διαδικασία όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Κατανοούμε την ανάγκη ή την, ε, το μέλημα επιτάχυνσης. Από την άλλη πλευρά, ε, από την πλευρά των εισηγητών βεβαίως ε, πρέπει να γίνει σεβαστό ένα χρονοδιάγραμμα και εμείς θα προσπαθήσουμε να το επιτύχουμε. Να θυμίσω ότι σήμερα το απόγευμα έχουμε κοινή συνάντηση με την ΑΦΚΟ θα έχουμε εκπροσώπους των Εθνικών Κοινοβουλίων επί του θέματος αυτού. Ε, σας καλώ λοιπόν να συμμετάσχετε και στη συνάντηση αυτή και όπως είπα θα προσπαθήσουμε να σεβαστούμε το χρονοδιάγραμμα. Αυτά και σας ευχαριστώ. Να περάσουμε στο επόμενο ή μάλλον όχι στο προηγούμενο θέμα. Αναγκαστήκαμε να το ε, τροποποιήσαμε. Αν η κυρία Άγγισε είναι ε, διαθέσιμη και είναι έτοιμη, παρακαλώ να της δώσω το λόγο. Thank you, uh, uh, uh, Chairman, and my apologies for my late arrival. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρησή μου. Θα αρχίσω με τα συμπεράσματα της έκθεσης. Θα ήθελα να σας πω ότι από τότε που επισκέφθηκε η αντιπροσωπεία μας τέλη Απριλίου επί τόπου υπήρχαν νέες εξελίξεις στην κατάσταση στην Καμπανία. Πρόσφατα η κατάσταση αποβλήτων στην περιοχή αυτή επιδεινώθηκε. Βλέπουμε δηλαδή να ε, επαναρχόμαστε στην κατάσταση που όπως ήταν πριν από μερικά χρόνια. Η κατάσταση ήταν πάρα πολύ άσχημη. Έγιναν διαδηλώσεις τις τελευταίες μέρες και μάθηκα για τον των ε, διαδηλώσεων αυτών υπήρχαν και τραυματίες. Αυτό καθιστά τη συζήτηση μας σήμερα πάρα πολύ επίκαιρη. Πρέπει να τονίσουμε αυτό, γιατί μπορούμε ίσως να επανέλθουμε κατά διάρκεια της συζήτησης. Είχαμε μια αντιπροσωπεία 7 μελών της Επιτροπής ε, Αναφορών και αυτό που είδαμε ήταν τέσσερα θέματα σημαντικά για να επιληθεί η κατάσταση. What apparently was missing. Αυτό που έλειπε ήταν ένα σχέδιο, ολοκληρωμένο σχέδιο για την <clears throat> επεξεργασία των πλήτων. Η... Συναντήσαμε τον κύριο Ρωμάνο. τον Υπουργό που ήταν αρμόδιος τότε και τώρα που έχει αναλάβει πλήρως το αξίωμά του. Είχε παρουσιάσει μια στρατηγική ε, που ήταν πάρα πολύ φιλόδοξη και που επικροτήθηκε από τα μέλη της αντιπροσωπείας μας. Αλλά βέβαια θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και κατά πόσο θα εφαρμοστεί το σχέδιο αυτό. Τι σημαίνει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο εξεργασία αποβλήτων. Αυτό σημαίνει ότι ο καλύτερος τρόπος είναι να αποφύγουμε τα αποβλήτα. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο. Εμείς δεν είδαμε όμως να υπάρχει μια ιεράρχηση των αποβλήτων στην καμπανία. Νομίζω ότι με την εφαρμογή ενός ε, σχεδίου που συμπεριλαμβάνει μια καλή ιεράρχηση θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Πρέπει βέβαια να υπάρχουν ε, οι λεπτομέρειες, να υπάρχουν τα benchmark, να υπάρχει δυνατότητα εποπτείας, να συλλέγονται στοιχεία. Συμπεριλαμβάνει επίσης την ε, στον καθαρισμό των περιοχών που έχουν ήδη μολυνθεί και στην ε, επίσκεψή μας στην ε, Καμανία είδαμε να υπάρχουν πολλές μολυσμένες περιοχές που πρέπει να καθαριστούν. Ε, σημαντικό είναι η συνεχής επιμόρφωση και πληροφόρηση και όσον αφορά τους αρμοδίους και όσον αφορά τους πολίτες. Είδαμε ότι εδώ και πολλά πολλά χρόνια ήταν υποδέκτης ε, ε, ε, αποβλήτων η καμπανία και εφόσον δεν μπορούν να τις τα δικά τους απόβλητα θα πρέπει να σταματήσουν αμέσως να δέχονται απόβλητα από άλλες περιφέρειες. Αυτό που λείπει από την όλη πολιτική και στην περιφέρεια είναι μια σχέση μεταξύ κυβέρνησης και πολιτών. Μια σχέση εμπιστοσύνης. Δεν υπάρχει κανένας διάλογος μεταξύ των πολιτών και της κυβέρνησης. Ίσως να άλλαξαν τα πράγματα εδώ μεταξύ. Α, αυτή όμως είναι η εικόνα που εμείς αποκομίσαμε τέλη Απριλίου. Και θα πρέπει να προσθέσω όπου τη φωσοφός των διαδηλώσεων που έγινε τώρα, χωρίς αυτό να είναι τα συμπεράσματα της αντιπροσωπείας, χρειάζεται, λέω, να συζητήσουμε την σχέση μεταξύ των αρχών και των πολιτών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι δεν θεωρείται πια ε, κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, αλλά παρόλα αυτά υπήρχε πολύ έντονη στρατιωτική παρουσία. Αλλά είπαμε βέβαια ότι η στρατιωτική επιτήρηση είναι αντίθετη προς την διαφάνεια, γιατί απαγορεύεται η πρόσβαση των πολιτών. Και αν θέλει κανένας να επαναφέρει την εμπιστοσύνη, θα πρέπει να ανοίξει τις ε, ε, τις, ε, τους χώρους αυτούς θα αφήσει και να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Πόρη τώρα. Είναι ένα θέμα που ζητήθηκε αναλυτικά μεταξύ των αρχών και της αντιπροσωπείας μας. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή, το, ο σωστός προπολογισμό που να χορηγηθεί από τις Ιταλικές, Κεντρικές και Περιφερειακές Αρχές. Υπάρχουν και κάποια χρήματα που έχει σταματήσει να έχει διακόψει την πληρωμή του η Κομισιόν, αλλά αυτό που προϋποθέτεται είναι η καμπανία να υποβάλει ένα σωστό πρόγραμμα και να αρχίσει και η επιτυχής εφαρμογή του. Και μόνο τότε θα μπορέσουν τα χρήματα αυτά από τα κοινωτικά ταμεία να επιλευθεθούν. Αυτό νομίζω ότι θα ήταν η σωστή άγουσα και διαδικασία. Υπάρχει τώρα βέβαια το βάρος του παρελθόντος. Όλα σκιάζονται από την κατάσταση, όπως σας είπα, κατεπήγοντος ε, μέχρι σήμερα. Αλλά όπως σας είπα, το θέμα είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα πρόγραμμα και η σωστή του εφαρμογή που θα βελτιώσει και τις σχέσεις κυβέρνησης πολιτών. Γιατί αυτή τη στιγμή η εμπιστοσύνη είναι τελείως στρεβλωμένη. Εμείς στην εταίρα, δεν είναι η, το θέμα της αντιπροσωπείας μας να αποφασίσει κατά πόσον η ατσέρα λειτουργεί σωστά ή όχι, αλλά το θέμα είναι ποια είναι τα στοιχεία, ποιο τα ελέγχει και κατά πόσο αντίθενται ελεύθερα στους πολίτες για να μπορούν να ελέγξουν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Καταλήξαμε επίσης στο συμπέρασμα ότι οι, οι χώροι των απορρίτων είναι κάτι που δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη. Ίσως θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν κάποια διαφορετική μέθοδος και όχι να ανοίγουν από εδώ και από εκεί ε, περιοχές ταφής. Αυτό που είναι ανα, απαράδεκτο είναι ότι στο Εθνικό Πάρκο του Βεζουβίου υπάρχει επίσης ένας χώρος ταφής, μου Τερζίνιο, που συνεχίζει, συνεχίζει να χρησιμοποιείται. Υπήρχε και... και υπήρχε και η Γκάβα, επίσης στο Εθνικό Πάρκο του Βεζουβίου, που επρόκειτο να, να ανοίξει, να αρχίσει να λειτουργεί. αλλά αυτή τη στιγμή ακούω ότι ο κύριος Περδουσκόνη χθε επιβεβαιώσει ότι αυτή, αυτός ο χώρος θα αφήσει δεν θα ανοίξει όπως μας είχαν υποσχεθεί όταν είμαστε στην Καβανία. Καλό είναι αυτό και ευχαριστώ από καρδιά στον κύριο ε, Μπερλουσκόνη γιατί μας το είχαν υποσχεθεί στην επίσκεψή μας και τελικά έγινε. Και ένα τελευταίο θέμα που θα ήθελα να σχολιάσω αυτή τη στιγμή είναι τα ειδικά απόβλητα και βιομηχανικά ε, απόβλητα. Μία αναφορά είχαμε σε αυτά και γι' αυτό δεν συγκεντρώσαμε την προσοχή μας κατά τη διάρκεια της ε, διαμονή μας στην ε, Καμπανία πάνω στο θέμα αυτό. Αλλά όμως ε, μας το είπαν αυτό εκεί γιατί είμαστε χώρα χώρο αφής του Τερζίνιο και μας είχαν πει ότι μόνο οικιακά απόβλητα ε, τα εκεί. Αλλά όταν πήγαμε επί τόπου είδαμε ξεκάθαρα ότι υπήρχαν και βιομηχανικά απόβλητα. Είναι απαράδεκτο να υπάρχουν σε αυτό το χώρο υγειονομικής ταφής ε, βιομηχανικά απόβλητα και είναι κάτι που θα πρέπει να εξεταστεί. Θα πρέπει οι αρχές να έχουν αυστηρό έλεγχο όσον αφορά την ε, αντιμετώπιση αυτών των ειδικών αποβλήτων. Και όλες οι αρχές, η κεντρική αρχή οι περιφερειακές αρχές, οι τοπικές αρχές θα πρέπει να σέβονται την κοινωτική νομοθεσία για τα απόβλητα. Τώρα, τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. θα πρέπει να κάνουμε. Είπαμε, η κυβέρνηση και οι τοπικέ αρχές θα πρέπει να έχουν ένα σωστό σχέδιο και να το αφαιρμάσουν και να είναι σύμφωνο και με την κοινωνική νομοθεσία. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την Ιταλία, να τη στείλουμε χείρα βοηθεία για να μπορέσει να μπορέσει να συμφορφωθεί με τον κοινοτικό νόμο. Η καμπανία από μόνη της προφανώς έχει δυσκολίες. Δεν έχει ολοκληρωθεί λοιπόν το θέμα. Θέλουμε να ενημερωθούμε, θέλουμε να ελέγχουμε την κατάσταση στην Ιταλία και θα ήθελα να προτείνω να παίξουμε ενεργό ρόλο στη διαδικασία αυτή. Να μην καταλήψουμε την, ε, αυτές τις αναφορές και να επανέλθουμε του χρόνου το 2011 ή αρχές του 2012 για να μπορέσουμε επιτόπου να ελέγξουμε τις εξελίξεις. Εδώ θα ήθελα να κλείσω την παρουσίαση αυτή. που σας ανέφερα τα σχόλια του Συνόλου της Αντιπροσωπείας και εγώ προσωπικά θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή Αναφορών να προωθήσει το θέμα αυτό στην Επιτροπή Περιβάλλοντος για να συζητηθεί εκεί. Όχι μόνο σχετικά με την Καμπανία, υπάρχουν πολλές περιοχές στην ε, Ευρώπη, ιδίως σε περιόδους οικονομικής κρίσης, που δεν έχουν είτε τους σπόρους είτε τις γνώσεις, είτε το, τους για να εφαρμόσουν ένα καλό πρόγραμμα. Θα ήθελα λοιπόν να στηρίξετε την ε, σύστασή μου, να συζητηθεί το θέμα αυτό στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και να περάσει για τον ίδιο λόγο και στην Ολομέλεια. Γιατί οι περιφέρειες με τις ε, δυσκολίες αυτές πρέπει να τύχουν της υποστήριξη και της βοήθειάς μας και θα πρέπει να συζητήσουμε πώς μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Τελειώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους που ήταν στην αντιπροσωπεία για τη θαυμάσια συνεργασία και να ευχαριστήσω και τους συνεργάτες μας που έπαιξαν τόσο σημαντικό ρόλο. Και όπως είπατε πρόκειται για πολύ καλή επίσκεψη. Είναι φεύγοντας είναι πιο σημαντική βέβαια. ήταν πάρα πολύ σημαντική κατά τη διάρκεια της ε, επίσκεψής μας. Και θα να πω ότι τύχαμε συνεργασία από τις αρχές και γι' αυτό προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας αυτής. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τη Νένφο Μέρκης και θα δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής, τον κύριο Μαγκανά. Καλή σας μέρα. Εκπροσωπώ εδώ την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, για να σας δώσω ε, μια επικαιροποίηση των ε, στοιχείων όσον αφορά την κατάσταση των απορριμμάτων στην Κατάνια. Όπως σας, Όπως σας είπα και στην προηγούμενη παρουσία μου στην Επιτροπή Μεταφορών, μετά από την απόφαση του δικαστηρίου, η Επιτροπή έστειλε επιστολή στις Ιταλικές Αρχές για να δουν μαζί τον τρόπο με τον οποίο θα έδινε οι τελικές αρχές συνέχιση ε, στο θέμα. Οι τελικές αρχές μας έστειλαν μία, ε, ε, ένα έγγραφο τον μήνα Ιούνιο, έγγραφο το οποίο αξιολογήθηκε από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αμέσως μετά τον Ιούλιο έλαβε χώρα μία συνάντηση με τις Ιταλικές Αρχές ακριβώς για να συζητηθεί το έγγραφο αυτό. Η Επιτροπή ζήτησε από τις Ιταλικές Αρχές να αποστείλουν ε, συμπληρωματική απάντηση γιατί το πρώτο έγγραφο θεωρήθηκε ανεπαρχές ε, μια και δεν ε, περιείχε αρκετά λεπτομερές χρονοδιάγραμμα. Ε, θέλαμε λοιπόν συγκεκριμένες ε, ε, ημερομηνίες για την υλοποίηση των εγκαταστάσεων. Πότε δηλαδή ε, προτίθεται οι, προτίθεται οι τελικές αρχές να κατασκευάσουν και να θέσουν σε ισχύ ε, τις ε, μονάδες. Επιβεβαιώθηκε η βούληση των Ιταλικών αρχών να θεσμοθετήσουν ειδικό πλαίσιο δράσης για την καμπάνια. Un progetto, un draft di ε, ένα ε, περιφερειακό πρόγραμμα λοιπόν ε, διαχείρισης το οποίο ζητήσαμε σαν υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μας υποβληθεί όσο γίνεται γρηγορότερα. Οι αρχές της καμπάνια θα επικεντρωθούν στο ότι το σχέδιο δράσης θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο, θα πρέπει να προβλέπει την ανακύκλωση την χρήση ε, όλων των ε, ε, ανακυκλώμενων υλικών. Και επίσης να υπάρξει ε, ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ε, ε, γρήγορη αποδόμηση του στόκ, το οποίο έχει δημιουργηθεί ήδη. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επίσης να υποβληθούν νέα προγράμματα διαχείρισης των απορριμμάτων γιατί πρέπει να σας πω ότι στην περιοχή υπήρχαν σχέδια ε, για τη διαχείριση των απορριμμάτων, αλλά δυστυχώς ποτέ δεν εφαρμόστηκαν. Επομένως, ε, η Επιτροπή ζητά όχι μόνο να υποβληθούν ε, τα προγράμματα και τα σχέδια, αλλά να υποβληθούν και όλα τα συνοδευτικά μέτρα τα οποία θα ληφθούν έτσι ώστε να λειτουργήσει σωστά όλο το σύστημα. Για να αξιολογηθεί το συμβατό ή όχι ε, της εγκατάστασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε επίσης να ε, εκπονηθεί μελέτη από εξωτερικό συνεργάτη. Επομένως, να αξιολογηθεί αυτό το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης ε, της καμπάνια από εξωτερικό μελετητή. Και τέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε επίσης από τις Ιταλικές Αρχές να προβλέψουν την δημιουργία μιας ιστοσελίδας όπου θα δημοσιευθεί, θα αναρτηθεί ε, αυτό το περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων έτσι ώστε και η Επιτροπή αλλά και οι πολίτες να μπορούν να παρακολουθούν ε, την ε, πρόοδο των εργασιών και την πρόοδο της υλοποίησης. Πρέπει να πω ότι κατά το παρελθόν εγκρίθηκαν πολλά ενδιαφέροντα και ικανοποιητικά περιφερειακά προγράμματα, τα οποία όμως δεν υλοποιήθηκαν σωστά. Ε, και προφανώς έτσι οδηγηθήκαμε στην ε, μεγάλη κρίση των ετών 2007-2008. Η Επιτροπή Ζητάει λοιπόν ενημέρωση, ζητάει επικαιροποίηση όλων των εγγράφων και των συμπληρωματικών εγγράφων και ζητά να ανακοινωθεί το νέο επικαιροποιημένο περιφερειακό πρόγραμμα διαχείρισης απορριμμάτων στη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος και βεβαίως θα αξιολογηθούν όλα τα έγγραφα αυτά όσο γίνεται γρηγορότερα έτσι ώστε να υπάρχει επιστροφή γνωμοδότησης προς τις Ιταλικές αρχές οι οποίες με τη σειρά τους θα μπορέσουν να προχωρήσουν στην υλοποίηση των προγραμμάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως πάντα, είναι ανοιχτή όσον αφορά τι εθνικέ αρχέ και κυρίαρχο στόχος είναι η επίτευξη λύση του εκάστοτε προβλήματος με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, με τον πιο αποτελεσματικό και γρήγορο τρόπο. Επομένως, η Επιτροπή κατά κάποιο τρόπο τίνει χείρα βοηθείας προς τις περιφερειακές αρχές ε, της ε, χώρας και τι εθνικέ ε, αρχέ και επομένως ε, θέλει να βοηθήσει και την περιφερειακή διοίκηση της Καμπανίας αλλά και την κεντρική Ιταλική κυβέρνηση. Ευχαριστούμε πολύ. Η συνάδελφοι Κοτσολίνη και Ριβελίνη μου ζήτησαν να πάρουν πρώτοι τον λόγο γιατί θέλουν να φύγουν. Ε, θέλετε να τους αφήσουμε να πάρουν τον λόγο πρώτοι. Όχι μάλλον, δεν ακούγεται η παρέμβαση της κυρίας Όκεν. Ε, να τους δώσουμε τον λόγο αλλά γρήγορα να μιλήσουν λίγο. Δεν θα μιλήσετε, ένα Κωνσταντίνο. Είναι σημαντικά τα νέα που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και βεβαίως θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την εργασία την οποία έχει εκπονήσει μαζί με την αντιπροσωπεία. Επίσης είναι γεγονός ότι ζούμε νέα ε, επίγουσα κατάσταση στην καμπάνια και επομένως ε, δικαιολογείται η προσοχή που δίνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Nelle prossime ore si giocherà una partita delicata θα παιχτεί ένα πολύ σημαντικό, ε, ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι ε, όσον αφορά το θέμα της χρήσης ε, των ε, εγκαταστάσεων γιατί μην ξεχνάμε ότι ε, το φυσικό πάρκο του Βεζούβιου είναι πολύ κοντά και εν πάση περιπτώσει είναι σημαντικό να έχουμε ένα περιφερειακό τοπικό σχέδιο, ένα πρόγραμμα περιφερειακό το οποίο θα είναι σφιχτό όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα. Γιατί ε, θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ε, ότι οι διάφορες αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν οπωσδήποτε θα έχουν επίπτωση ε, στην εμπορική, οικονομική ζωή, στη ζωή των πολιτών. Και βεβαίως να μην ξεχνούμε ότι ε, πέρα από κάθε ε, ιδιαίτερα σύγχρονο και καινοτόμο σχεδιασμό ε, ή μάλλον πίσω από κάθε σύγχρονο και καινοτόμο σχεδιασμό ελοχεύει το πρόβλημα της χρηματοδότησης. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξει και η, η χρηματοδότηση αυτή. Και βεβαίω θέλουμε και η Επιτροπή ε, Περιβάλλοντος και η, Επιτροπή, η Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος Επιτροπής να μην ασχοληθούν με το θέμα μόνο και επικεντρωμένα με την, με το, με την ε, υπόθεση της καμπανία, αλλά και γενικότερα όσον αφορά αυτό το ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ο συνάδελφος Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω εκείνους που οργάνωσαν τα ταξίδι την Επιτροπή και τους Ιταλούς ε, ε, συναδέλφους και την Πρόεδρο που μας έδωσε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες επί τόπου. Η αποστολή αυτή ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και πλήρες. Δεν είχαμε καθόλου χρόνο να βαρεθούμε ούτε τίποτα. Εγώ πολλά έμαθα. με διάφορα προβλήματα. Ε, εγώ είχα τρία προβλήματα που αφορούσαν την ε, νομική πτυχή, που αφορούσαν τα βιομηχανικά απόβλητα όπου υπάρχει από ό,τι φαίνεται παράνομη ταφή και είχαμε το πρόβλημα με γενικά παράνομες, ε, παράνομους χώρους ε, μάλλον των απορρίτων. Αν μπορέσουμε από κοινού με τις αρχές και τους πολίτες της καμπανίας και με τους εκπροσώπους της Επιτροπής να λύσουμε τα προβλήματα για τα τις νόμιμες, ε, τους νόμους χωροσταφείς θα μπορέσουμε μετά να λύσουμε και το θέμα των παράνομων. Ακούγεται ε, κάπως αντίστροφο, αλλά είναι σωστή μέθοδος. Μετά θέλω να πω ότι όταν έχουμε διάλογο με τους πολίτες θα πρέπει η κύρια μας περίμενα να είναι η διαφάνεια. Γιατί αλλιώς ε, ο άλλο, η μεν λένε το ένα, η δεν λένε το άλλο και δεν υπάρχουν στοιχεία. Και αυτό που χρειάζεται είναι ακριβώς να υπάρχουν στοιχεία καταμέτρησης. Δεν μπορέσει να υπάρχει και ανταλλαγή των απόψεων αυτών μετά. Επικοδομητικό διάλογο. Το πρόβλημα που βλέπω και εδώ είναι μια ερώτηση προ την Κομισιόν. Είναι το εξή. Λέμε ότι χρειαζόμαστε βέβαια ιδέε και σχέδια σωστά και βάσιμα για να μπορέσουμε να δώσουμε τα χρήματα. Πρώτη ερώτηση. Τι χρονικό ορίζοντα βλέπει η Κομισιόν εδώ. Πότε θα απελευθερωθούν τα χρήματα αυτά δηλαδή από εκεί και πέρα. Κατόπιν. Μπορούμε να αναπτύξουμε μια διαδικασία βήμα προς βήμα σαν κατεπίγουσα βοήθεια. Ε, τώρα να πω, οι παλιές, ε, οι παλιοί χώροι ταφής έχουν γεμίσει. Καινούργοι χώροι υγειονομικής ταφής ή δεν γίνονται ή θα πρέπει να του ανηθούμε για λόγου προστασία του περιβάλλοντο. Πραγματικά πολλέ φορέ μα όκαρε το γεγονό σε τι καταπληκτικά τοπία τοποθετούν τη, τους χώρους αυτούς Λοιπόν, ίσως θα πρέπει να υπάρχουν και εκτεφρωτές. Και αν υπάρχει μια γενική, ένα γενικό σχέδιο σωστό, δεν θα μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε βήμα προς βήμα. Γιατί εγώ φοβούμαι ότι συζητάμε και ξανασυζητάμε τα σχέδια και τα προγράμματα και σε λίγο θα έχουμε την ίδια κατάσταση που είχαμε και στο παρελθόν, μια που έχουν γεμίσει οι νόμιμοι χώροι ταφή. Και την επόμενη φορά φαντάζομαι η καταστροφή θα είναι ακόμα πιο έντονη από την προηγούμενη φορά. Γιατί δεν θα έχουν καμία κατανόηση πια οι πολίτε. Ρωτώ την Κομισιόν πώ μπορούμε να έχουμε μια διαδικασία βήμα προ βήμα που να χρηματοδοτεί και επιμέρου ε, επιμέρους ε, σχέδια να μην περιμένουμε χρόνια και χρόνια και να επιδεινωθεί η κατάσταση. Ευχαριστώ. Η κυρία Ευχαριστώ. Φυσικά και συμφωνώ με τους συναδέρφους και ευχαριστώ για την ε, τόσο καλή συνεργασία. Θέλω όμως να τονίσω μερικά ζητήματα. Αυτή η συνεχιζόμενη χρήση του κατεπήγοντος. Όταν έχουμε ερωτήσεις. Σύμφωνα με τον Ιταλικό νόμο, είναι νόμιμο. Ποιος ήτανε. Ντέλα Μασέριο. Ήμασταν εκεί, σε ένα πολύ ωραίο μέρος. Και μετά αποδείχθηκε χωματερή. που απειλούσε το νερό, τα πάντα. Και με το κατεπήγον δηλαδή γίνεται. Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα. Πρέπει λοιπόν στο μέλλον να τονίσουμε ότι σεβόμαστε τους πολίτες όταν θεωρούν εγκληματίες αυτούς που διαμαρτύρονται για κάτι τέτοιο, οι κυβερνήσεις τους θεωρούν δηλαδή εγκληματίες, εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορεί να θεωρούνται αυτοί οι κακοί επειδή διαμαρτύρονται για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να φροντίσει όταν έχουμε ένα σχέδιο να ξέρουμε ότι είναι πραγματικότητα. Γιατί από σχέδιο άλλο τίποτα το πώς πρέπει να είναι. Η πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική συχνά. Να βλέπουμε ότι είναι σύμφωνο το σχέδιο με το αποτέλεσμα. Και αναφερόμαστε καμιά φορά στη Δανία και για τις μονάδες καύσης που έχουμε εκεί. Εμείς έχουμε μάθει ότι δεν φτάνει να διαθέτει κανείς την υπέροχη τεχνολογία. Αν έχεις χημικά, ηλεκτρονικά απόβλητα, δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη στάχτη. Πρέπει να είναι καθαρή η στάχτη για να μπορεί μετά να ανακυκλωθεί και να χρησιμοποιηθεί η στάχτη αυτή. Αν είναι από χημικά δεν μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις μετά τη στάχτη από την καύση. Μας είπαν επίσης ότι η λειτουργία της μονάδας είναι πολύ απαιτητική. Δεν γίνεται ο έλεγχος έτσι εύκολα. Υπάρχουν προβλήματα με τις εκπομπές. Εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά. και βλέπουμε ότι πάνε οι στρατιώτες και προσπαθούν να διώξουν τον κόσμο, να μην πλησιάσει ο κόσμος. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με την απειλή αυτή λοιπόν. Το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί αν δεν συμμετέχουν και οι πολίτες. πρέπει να υπάρχει σεβασμός λοιπόν για τους πολίτες. Και οι πολίτες βέβαια πρέπει να σέβονται τις αρχές. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο και στο μέλλον και ζητάω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να το φροντίσει αυτό. Αλλιώς ξεχάστε το. Επίσης θέλω να πω για τον συνάδελφο Πίτερ Γιάρ. Δεν κοιτάξαμε πραγματικά βιομηχανικά απόβλητα. Έχω την αίσθηση, δεν ξέρω, αλλά νομίζω ότι η πραγματική προβληματική είναι οι βιομηχανίες. Ίσως μεθαύριο ασχολούμαστε μόνο με τις υποδομές. Θέλουμε να κοιτάξουμε τις υποδομές που θα εξυπηρετήσουν τη βιομηχανία σε μια περιοχή κλπ. Ωραία. Αλλά πρέπει επίσης να επικεντρωνόμαστε και σε κάτι άλλο, στο τι γίνεται μετά. Γιατί και στη Γερμανία και αλλού διαπιστώνουμε ότι τα βιομηχανικά απόβλητα τελικά καταλήγουν σε αυτούς τους χώρους που δεν θα έπρεπε. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Ντεμπρούν. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μάκης για την τόσο ξεκάθαρη παρουσίαση που μας κάνατε της επίσκεψης αυτής. Πάλι η σημερινή συζήτηση ήταν πολύ καλή για αυτή την τόσο δυσάρεστη κατάσταση. Το είπε και την προηγούμενη φορά που το συζητήσαμε εδώ, ότι η κατάσταση είναι από εντελώς απαράδεκτη έως απαράδεκτη. Πρέπει να το καταλάβουμε ότι μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο συζητάμε. Ξέρω ότι περνάει ο χρόνος, οπότε μερικές ερωτήσεις πρώτα απ' όλα. Η κυρία Μάκης μίλησε για την δυσκολία που υπάρχει για τη συλλογή πληροφοριών, διάλογο κτλ. μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης. Θα μπορούσατε να δεχτείτε μια προφορική τροπολογία να τη συμπεριλάβετε στην έκθεση που να λέει το εξή. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, τον κύριο Τομασίτου, οι πολίτες δεν έχουν πρόσβαση σε διάφανη και ξεκάθαρη ενημέρωση ούτε μπορούν να συμμετέχουν στην αξιολόγηση των κινδύνων για το περιβάλλον και την υγεία, όπως φάνηκε στην περίπτωση της μονάδας ε, καύσης στην Ατσέρα. Θα θέλατε να δεχτείτε αυτή την ε, προφορική τροπολογία. Εισηγήτρια, στρέφομαι προς τους άλλους. Από τη στιγμή που λέει ότι είναι ο δήμαρχος που το λέει αυτό, για μένα δεν υπάρχει πρόβλημα. Πρόεδρος. Συνεχίζει η συγκήτρια. Για μένα είναι αποδεχτή αυτή η τροπολογία. Το πρόβλημα είναι ότι αν δεχτώ την ε, προφορική τροπολογία ε, θα μου τραβήξει μετά το αυτή η γραμματεία μου. Δηλαδή η προφορική τροπολογία θα πρέπει να υποβληθεί, να γίνει σαφής ε, η αποδοχή από τις ε, ε, ομάδες και επίσης και η ίδια η εισηγήτρια να δει εάν δέχεται την τροπολογία αυτή. Δηλαδή υπάρχει ένα ζήτημα για το κατά πόσον είναι ανοιχτό το, είναι αποδεκτό συγγνώμη, το περιεχόμενο της προφορικής τροπολογίας. μέχρι να λήξει αυτό το διαδικαστικό θα δώσω τον λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να απαντήσει σε αυτά που είπαμε τώρα. Η κυρία Τεπρά, να συνεχίσω και με τα άλλα σημεία που είχα, γιατί δεν είχα μόνο αυτό. Α, νόμιζα ότι είχατε τελειώσει, λέει ο Πρόεδρος, επειδή πήρε το λόγο μετά η κυρία Μέρκης, αλλά παρακαλώ, συνεχίστε. Τεπρά. Δύο άλλα σημεία ήθελα να θίξω. Το ένα Μάλλον κανένα δεν υπάρχει στο κείμενο, αλλά επειδή αναφέρθηκε η κυρία Μάκης, είπε ότι δεν έχει κλείσει υπόθεση, ότι πρέπει να συνεχίσουμε να ενημερωνόμαστε κτλ. Και επειδή όλε οι αναφορέ που υπάρχουν για αυτό το θέμα πρέπει να παραμείνουν ανοιχτέ και να συνεχίσει η ενημέρωση, να σα πω ότι συμφωνώ απόλυτα και έπειτα το συζήτησα και με την Επιτροπή και θα το ξανασυζητήσω. Άκουσα ότι έχει αναλυφθεί δέσμευση όσον αφορά την καμπάνια, ότι, την καμπανία, ότι η περιφέρεια θα αγοράσει 252 ε, εκατομμύρια, κάτι Και μερικά από τα χρήματα αυτά είναι κοινοτικά. Θέλω λοιπόν να το ελέγξω. Ισχύει κάτι τέτοιο. Σκοπεύουν να αγοράσουν την μονάδα Και στέκει αυτό. Βάσει της δικιάς μας οδηγίας ε, για τα απόβλητα γίνεται κάτι τέτοιο, συνάδει. Grazie, Ωραία, θα ξαναδώσω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Παρακαλώ. Εάν κατάλαβα καλά την ερώτηση του κυρίου Γιάρα, δηλαδή υπάρχει κίνδυνος στην επικαιροποίηση του νέου ε, προγράμματος διαχείρισης, του νέου σχεδίου διαχείρισης, και αναμένοντας αυτό το μεγάλο ας πούμε σχέδιο διαχείρισης ε, να μην ε, γίνει τίποτα και επομένως να φτάσουμε σιγά σιγά ε, σε μια, ξανά, σε μια νέα μεγάλη κρίση. Βεβαίω πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα εξεκολουθήσει να ασκεί πιέσει και να επιμένει στι Ιταλικέ Αρχέ έτσι ώστε να λαμβάνονται σιγά σιγά τα μέτρα μέχρι να αρχίσει να ισχύει το ε, πιο σημαντικό σχέδιο. Υπάρχουν επίσης ε, κάποια προγράμματα τα οποία πρέπει να αρχίσουν ήδη. Ε, δηλαδή δεν θα περιμένουμε το νέο περιφερειακό σχέδιο διαχείρισης για να ξεκινήσει η οικοδόμηση των νέων εγκαταστάσεων που έχουν ήδη προβλεφθεί. αλλά μας λείπουν ακόμα στοιχεία. Δεν έχουμε στοιχεία για τα απόβλητα τα οποία έχουν συσσωρευμένα οι διάφορες χωματερές, αλλά σίγουρα θα χρειαστούν γύρω στα δύο χρόνια μέχρι να ομαλοποιηθεί ε, το πρόβλημα. Και οπωσδήποτε σε αυτά τα δύο-δυόμιση χρόνια θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, μην επαναληφθεί μια μεγάλη κρίση σαν αυτή του 2007 όσον αφορά τώρα την ιεράρχηση. Στο νέο πρόγραμμα διαχείρισης της ε, καμπανίας οι Ιταλικές αρχές έχουν δεσμευτεί να εγκρίνουν λοιπόν ένα ε, σχέδιο το οποίο θα σέβεται τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και εν πάση περιπτώσει το σχέδιο αυτό θα υποβληθεί στην ε, Κομισιόν η οποία θα πάρει και τις τελικές αποφάσεις. Επανειλημμένα έχει πει η Κομισιόν ότι μία από τις ε, προϋποθέσεις έτσι ώστε να ε, δοθούν τα, οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι να ευθυγραμμίζονται τα προβλεπόμενα στο σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων της καμπανίας με το πλαίσιο πλαίσιο διαχείριση απορριμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά τώρα την διαφάνεια, βεβαίω και αυτό το είπαμε ε, και το καταστήσαμε σαφέ ε, στι ιταλικέ αρχέ. Είπα και στην πρώτη μου παρέμβαση ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από τις Ιταλικές αρχές ε, να δημιουργήσουν μία ιστοσελίδα όπου και θα δημοσιευθεί ε, το νέο πρόγραμμα διαχείρισης και θα δημοσιεύονται οι εκάστοτε επικαιροποιήσεις και θα μπορούν και οι πολίτες ε, να κάνουν τα σχόλιά τους. Μέχρι τώρα οι απαντήσεις και η ανταπόκριση που είχαμε ήταν θετική γιατί ήδη στην ιστοσελίδα της περιφέρειας ε, της ε, Καμπανίας τέλη Αυγούστου αναρτήθηκε ένα έγγραφο το οποίο δεν είναι το τελικό, δεν είναι αυτό καθεαυτό ε, το σχέδιο διαχείρισης, αλλά είναι ένα προγραμματικό έγγραφο το οποίο αναφέρεται στον σχεδιασμό σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ε, αναρτήθηκε για δημόσια διαβούλευση επί 45 ημέρες. Contiene degli orientamenti ancora abbastanza generali. Ε, και επομένως ήδη είναι ένα πρώτο βήμα προς τη διαφάνεια και ένα βήμα βεβαίως προς την πληροφόρηση, προς την διαβούλευση με τους ε, πολίτες. Ελπίζω να απήντησα στις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ακόμα προσπαθούμε να λύσουμε από τεχνικής και ε, ε, έτσι, ε, διαδικαστικής απόψεως το ζήτημα που πρότεινε η κυρία Ντεμπρόν. Θα ήθελα και εγώ να κάνω κάποιες σκέψεις. Πιστεύω ότι η έκθεση της συναδέλφου Μέρκες σαφέστατα είναι καρπός ενδελεχούς και προσεκτικής εργασίας ε, στην οποία συμμετέσχουν και πολλοί συνάδελφοι και είμαι πολύ ευτυχής ε, που είδα πολλοί συνάδελφοι να ασχολούνται με ένα ζήτημα το οποίο και λόγω του ότι ε, προέρχομαι από αυτήν την ε, περιοχή ε, με συγκινεί ιδιαιτέρως και βεβαίως με κάνει κατά κάποιο τρόπο και ενεργητικά συμμετέχουσα αλλά και παθητικά δεχόμενη της πρωτοβουλίες που αφορούν αυτήν την περιφέρεια θα ήθελα να πω δύο-τρία λόγια μονάχα, να κάνω δύο-τρία σκέψεις, να τις υποβάλω στους ε, συναδέλφους εάν θέλουν ε, να τις χρησιμοποιήσουν. Στην έκθεση, μάλλον στον πρόλογο, η συνάδελφος Μέρκης, πριν από την ίδια την ε, έκθεση, έκανε κάποιες γενικές θεωρήσεις επί της παρούσης καταστάσεως. Ε, από τη στιγμή που έγιναν διάφορες ταραχές τις τελευταίες εβδομάδες ε, θα ήθελα να πω ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι επιδεινώθηκε η κατάσταση. Η κατάσταση είναι η ίδια, ε, αυτή την, την οποία δυστυχώς διαπιστώσαμε και εμείς τον Απρίλιο όταν επισκεφθήκαμε την περιοχή. Είναι μια κατάσταση δύσκολη και ε, όπως και ο κύριος Ρωμάνο μας είπε στη συνάντηση που είχαμε και εδώ στις Βρυξέλλες είναι μια ε, ε, κατάσταση δύσκολη από τη στιγμή που καταλαβαίνουμε ότι πέρα από τα καινούργια απορρίμματα υπάρχουν και αυτά τα στόκ των απορριμμάτων τα οποία κάποια στιγμή ε, με κάποιο τρόπο θα πρέπει ε, να ε, λυθούν αλλά βεβαίως αυτό δεν μπορεί να γίνει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Υπάρχει επίσης ένα έγγραφο το οποίο ατύπως ε, ε, μας ε, έχει δώσει η Δημαρχία της Νάπολης. Υπάρχουν κάποιες εξελίξεις οι οποίες αφορούν όμως μονάχα την Νάπολη, μονάχα την πόλη δηλαδή της Νάπολης είναι ένα πρόβλημα το οποίο αφορά έλλειψη οικονομικών πόρων ε, και σαν αποτέλεσμα είχε να σταματήσει η περισυλλογή των σκουπιδιών στην πόλη της Νάπολης. Υπήρξε μια, ένα λαϊκό κίνημα το οποίο σιγά σιγά πήγε και σε άλλες ε, περιοχές ε, γιατί όπως είπε και ο συνάδελφος Γιάρα και άλλοι συνάδελφοι δυστυχώς οι πολίτες ε, μετά από τόσα προβλήματα επί τόσα χρόνια ε, ε, ζουν μέσα σε μια κατάσταση τρομακτικής ανησυχίας και ακόμα και με το παραμικρό ξεσηκώνονται γιατί πραγματικά τους πιάνει πανικός και τρόμος. η Νάπολη και η Καζέρτα μονάχα ζήτησαν, την, ε, ε, τη, ζήτησαν νέα προγράμματα ε, στις άλλες ε, περιφέρειες ε, υπάρχει μια ομαλοποίηση. Η Νάπολη και η Καζέρτα παρουσιάζουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Έχουν ένα και μόνο όμιλο που ασχολείται με την συγκομιδή των σκουπιδιών και επομένως εδώ δυσκολεύεται λίγο η κατάσταση. Επίσης, η έλλειψη πόρων οδήγησε σε στάση πληρωμών των ε, ε, ε, ασχολούμενων με την καθαριότητα και επομένως γίνεται μία προσπάθεια απελευθέρωσης πόρων από την κεντρική κυβέρνηση, από τη Ρώμη, έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί ε, η ε, συγκομιδή των σκουπιδιών. Ε, όμως η Κομισιόν δέσμευσε τους πόρους γιατί δεν υπήρξε πλήρωση των προϋποθέσεων σε περιφερειακό τοπικό επίπεδο. Αλλά νομίζω ότι έτσι όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση θα επιτευχθεί τελικά από πλευράς της πόλεως της Νεαπόλεως η απεμπλοκή της κατάστασης και επομένως να ε, υπάρξουν ε, τα χρήματα αυτά διαθέσιμα. Επίσης, ε, όπως ανέφερε και η κυρία Μέρκης προηγουμένως, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Μπερλουσκόνη ανακοίνωσε το άνοιγμα ενός δεύτερου χώρου ταφής απορριμμάτων και επομένως αυτό οπωσδήποτε θα βοηθήσει. Αυτό μας το είχε ήδη προαναφέρει ο νεοεκλεγής ε, περιφερειάρχης. Επίσης ε, ο, ο κύριος Ρωμάνο ε, μας είπε ότι δεν θα υπάρξει δεύτερη χωματερή στο Καγιάνο. Όλα αυτά και η στρατηγική την οποία ε, ε, προβλέπει η περιφέρεια ε, έχουν κοινοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Προβλέπεται συγκεκριμένα η υποβολή νέου σχεδίου, βεβαίως η οποία θα ακολουθείται από προσχέδιο χρονοδιαγράμματος. Συζητήθηκε το θέμα αυτό με την Επιτροπή. Όπως είπα και προηγουμένως, οι περιφέρειες έχουν ε, υποβάλει τα προγράμματά τους, τρεις μεταξύ αυτών. Οι άλλες δύο που ανέφερα και προηγουμένως αναμένεται να το πράξουν σύντομα. Ε, τα ε, όσα μας είχε ανακοινώσει ο κύριος Ρωμάνο όταν ήρθε εδώ στις Βρυξέλλες έχουν ήδη ε, εγκριθεί από το Δημοτικό και Περιφερειακό Συμβούλιο. Επίσης ε, το σχέδιο προστασίας του, της ποιότητας του αέρα και το σχέδιο παρακολούθησης του περιβάλλοντος και, της, συγγνώμη, των υδάτων ήδη είναι έτοιμα για συζήτηση. Και όπως όπως ε, μας είπε και ο κύριος ε, Ρωμάνο, ε, μέχρι την 31η Δεκάτου του 2010 θα έχουν ολοκληρωθεί τα σχέδια αυτά και θα αρχίσουν να υλοποιούνται. Όσον αφορά τώρα την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ε, θα ολοκληρωθεί την 31η ε, ε, Δεκεμβρίου του 2010 και όπως μας είπε και ο κύριος Ρωμάνο και εδώ πρέπει να πω ότι διαβάζω τα πρακτικά έτσι όπως μας τα έχουν δώσει υπάρχουν κάποιες υπάρχουν ακόμα κάποιες γραφειοκρατικές κατά κάποιο τρόπο δομές οι οποίες ακόμα υπάρχουν και που είναι απόρρια της νομικής κατάστασης εκτάκτου ανάγκης και αυτές θα λειτουργήσουν μέχρι τον Ιανουάριο του 2011 επανειλημμένα ε, συζητήθηκε και μας το τόνισε και ο ε, Σύμβουλος ότι θα πρέπει να ε, συζητηθεί και έχει ξεκινήσει ήδη μία συζήτηση με τοπικούς φορείς για την δημιουργία μερικών ε, ε, χωματερών ακόμα που όμως ε, η τοποθεσία τους θα επιλεγεί με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στον υδάτινο ορίζοντα της περιοχής. Όσον αφορά τώρα τις λοιπές δραστηριότητες, ε, πρέπει να πω ότι για την ε, Ανατολική Ναπολή το θερμοηλεκτρικό, ε, η θερμοηλεκτρική μονάδα καύσης έχει ήδη προχωρήσει πάντα μέσα στο πρόγραμμα πλαίσιο προστασίας των εδαφών και του υπεδάφους του Περιφερειακού Συμβουλίου της Νάπολης και βρίσκεται ήδη σε επίπεδο προμήθειας για την περιφέρεια του Σαλέρνο υπήρξε μια ε, ισχυρή αντιπαράθεση μεταξύ κοινοτικής, τοπικής διοίκησης και κεντρικής διοίκησης όσον αφορά ε, τον ορισμό συμφωνίας ε, ανάμεσα στις δύο πλευρές. Έχει και εκεί ξεκινήσει σιγά σιγά η διαδικασία και έχει ξεκινήσει ήδη η δεύτερη, η δεύτερη προκήρυξη. Όσον αφορά τώρα τις, τις μονάδες επεξεργασίας σκουπιδιών στην Δυτική Νάπολη. Αυτό θα αρχίσει να ισχύει από την επόμενη χρονιά. Ε, παραπάνω από 80.000 τόνοι ε, οργανικών σκουπιδιών ε, θα μπορέσουν να ε, περάσουν ετησίως από τη μονάδα αυτή. Τώρα ενδεχομένως αν θέλετε κάποια άλλα στοιχεία θα μπορούσαμε να τα βρούμε. Εν πάση περιπτώσει εγώ ανεπισήμως μπορώ να σας δώσω και όλα τα έγγραφα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Και να πω επίσης ότι μέσω των μονάδων καύσης θα μπορέσουμε σιγά σιγά να ε, ε, αντιμετωπίσουμε το ήδη συσσωρευμένο στόκ των σκουπιδιών. Ε, κοιτάξτε, οι πολίτες πλέον απαιτούν λύση και εμείς είμαστε εδώ έτσι ώστε να βρούμε όσο γίνεται καλύτερα πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα αιτήματα, τα πιεστικά πλέον αιτήματα των πολιτών. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Πρέπει να πω ότι εδώ και δύο χρόνια λειτουργεί και ένα τηλεφωνικό ε, κέντρο όπου μπορούν οι πολίτες ε, να ενημερώνονται. Επίσης έχει ανοίξει ε, και ένα πόρταλ στο οποίο μπορούν οι πολίτες να ενημερωθούν για όλα τα επίσημα έγγραφα τα οποία σχετίζονται με το θέμα τους και τα οποία έχουν κυκλοφορήσει Τέλος, να σας πω ότι συνεχίζουν όλες οι συζητήσεις, οι ανοιχτές συζητήσεις με τους ε, πολίτες μέσα από ένα βεβαίως δημοκρατικό και αντιπροσωπευτικό ε, σύστημα, μέσα ε, από τα διάφορα όργανα, τους αιρετούς λοιπά της περιοχής. Ήθελα να τα προσθέσω αυτά που σας είπα ακριβώς για να καταλάβετε ότι γίνονται ε, κάποια, κάποιες κινήσεις εμείς στην Κομισιόν ή στο Κοινοβούλιο. Βεβαίως δεν έχουμε στα χέρια μας όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα μας επιτρέψουν να λύσουμε αυτό το δραματικό ζήτημα. Αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να βοηθήσουμε ή μπορούμε ε, να πιέσουμε έτσι ώστε να ε, πιέσουμε για να επιταχυνθούν οι χρόνοι και όπως ε, ε, πολύ ειλικρινά δέχτηκε ο ε, κύριος Ρωμάνο όταν τον συναντήσαμε είναι γεγονός ότι τα προβλήματα έχουν συσσωρευτεί, έχουν συσσωρευτεί και από προηγούμενες διοικήσεις αλλά αυτή τη στιγμή λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα υπό την προσεκτική ματιά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Να σας πω επίσης ότι έγινε η τελική περαίωση για το, από το Διοικητικό Δημοτικό Συμβούλιο και Περιφερειακό Συμβούλιο για τα έτη 2007-2000-2007 και επομένως ε, ε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν ε, περίπου 350 εκατομμύρια ευρώ τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για, την, για τον νέο σχεδιασμό, το νέο περιφερειακό σχέδιο για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Βεβαίως ε, ε, ε, η περιφέρεια προτίθεται να προχωρήσει αν και εάν βοηθήσουμε και εμείς ενδεχομένως οι χρόνοι θα επιταχυνθούν έτσι ώστε να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτός ο τόσο σημαντικός σχεδιασμός που πραγματικά είναι η προσμονή όλων των πολιτών. Μου λέει η γραμματεία ότι όσον αφορά το αίτημα προφορικού ε, προφορικής τροπολογίας ε, ε, η συνάδελφος την απέσυρε γιατί υπάρχει ήδη η τροπολογία το περιεχόμενο αυτής της προφορικής τροπολογίας υπάρχει ήδη στην Ολομέλεια στην έκθεση συγγνώμη όχι, είναι επειδή μου είπαν ότι είναι τεράστιο μπελά και καλύτερα να μην το κάνω. Γι' αυτό. Ευχαριστώ. Δεν είχα καταλάβει καλά, μου έδωσαν λάθο πληροφόρηση, λέει η Πρόεδρο. Πάρα πολύ ωραία. Θα καταγραφεί έτσι κι αλλιώ στα πρακτικά το έτοιμά σα. Πρέπει τώρα να ε, περάσουμε στην έγκριση του εγγράφου. Μια και δεν είναι επίσημη ψηφοφορία. Απλώς θέλω να μου πείτε εάν υπάρχουν κάποιες ψήφοι εναντίον ή κάποιες αποχές. Όχι, δεν βλέπω να καταψηφίζει κανείς την έκθεση αυτή. Ε, εγώ λαμβάνοντας υπόψη την προσωπική ας πούμε σχέση θα ήθελα να ε, δηλώσω ότι ψηφίζω αποχή. και θα ήθελα να ζητήσω από την ε, επικεφαλή της αντιπροσωπείας, την κυρία Μέρκης, να... Ε, ε, μάλλον θα μεταφέρω έτοιμα και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος έτσι ώστε τέτοιου είδους κρίσεις που προκαλούνται λόγω των σκουπιδιών, λόγω των απορριμμάτων να φτάνουν στην Ολομέλεια. Ωραία. Ε, όσον αφορά αυτή την σύσταση προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος, ποια είναι η θέση υπέρ από ό,τι καταλαβαίνω, υπέρ είναι όλοι οι συνάδελφοι. Πάρα πολύ ωραία, επομένως εμείς ε, θα κάνουμε την εν λόγω σύσταση στην Επιτροπή Περιβάλλοντος. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποιον άλλον που ζητάει το λόγο. Η συγγήτρια. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Ναι, Κατάλαβα ότι θα περάσουμε μέσω της Επιτροπής Περιβάλλοντος για να πάμε στην Ολομέλεια, σωστά. Δηλαδή μαζί με το περιβάλλον θα πάμε στην Ολομέλεια για να το συζητήσουμε και να γίνει εκεί η γενική συζήτηση, σωστά. Πρόεδρος, ναι, ναι. Θα κάνουμε ένα αίτημα, σύσταση μάλλον, προς την Επιτροπή Περιβάλλοντος και η Επιτροπή Περιβάλλοντος θα φέρει το θέμα στην Ολομέλεια. Κύριος Γιάρ για το ίδιο θέμα. Ναι. Όλα σωστά. Είπαμε ότι δεν πρέπει μόνο για την καμπανία. Πρόκειται γενικά για την ε, εξαρτησία απορριμμάτων στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να προτρέχουμε βέβαια την απόφαση της Επιτροπής Περιβάλλοντος. Θα πρέπει να είμαστε δικαίοι των συναδέλφου τη και να μην προδικάζουμε την απόφασή του. Ε, Ωραία, λέει η Πρόεδρο. Εμεί θα προτείνουμε το θέμα στην επόμενη συνάντηση των συντονιστών. Ενδεχομένω θα καλέσουμε την κυρία Μέρκη έτσι ώστε να ασχοληθεί προσωπικά και με το ε, θέμα αυτό. Και μετά στους συντονιστές θα καθορίσουμε τις λεπτομέρειες της διαδικασίας. Σας ευχαριστώ όλους και περνάουμε λοιπόν στο επόμενο σημείο. Eh, Ο David Law μου λέει να σας προτείνω και εδώ μία περαιτέρω αντιστροφή. Έχουμε το τελευταίο σημείο της ημερήσιας διάταξης για το οποίο είναι εδώ οι αναφέροντες. Ενώ ε, τα σημεία 19 και 20 δεν έχουν παρουσία των ε, ε, των ε, αναφερόντων, επομένως να περάσουμε άμεσα στην, ε, στην 417 του 2009 και θα δώσω τον λόγο στον κύριο Ντάμπρα. Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, είναι μεγάλη μου τιμή που ε, με δέχεστε εδώ και με προτίθεστε να ακούσετε τη γνώμη μου εδώ στην Επιτροπή ε, σας ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και εκπροσωπώ βεβαίως εδώ χιλιάδες Ευρωπαίους πολίτες. Η πρωτοβουλία ξεκινάει από το άγχος το οποίο αντιμετωπίζουμε όσον αφορά την αποτυχία των Ιταλικών θεσμών να νομοθετήσει σε σχέση με μια λαϊκή πρωτοβουλία η οποία προβλέπεται από το Ιταλικό Σύνταγμα και το οποίο έχει υπογραφεί από πάνω από 35.000 πολίτες την 8η Σεπτεμβρίου 2007 και η οποία προβλέπει απαγόρευση εκλογής σε καταδικασμένους. Έχουν περάσει τρία χρόνια και αυτός ο νόμος ακόμα βρίσκεται ε, στο ψυγείο της ε, Ιταλικής ε, Γερουσίας. Γιατί οι βουλευτές οι οποίοι δεν εκλέγονται από τους πολίτες αλλά μονάχα από τις λίστες των κομμάτων τους έχουν άλλα πράγματα να κάνουν, όπως ας πούμε να περάσουν τον ε, αντισυνταγματικό νόμο Λόντο Αλφάνο που προέβλεπε δικαστική ασπίδα προστασίας για τον Πρωθυπουργό και που εγκρίθηκε αμέσω μέσα σε 10 μέρες μετά από την πρώτη συζήτηση και που βεβαίως παρότι ε, υπεγράφει αμέσω από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ε, τελικά ανεστάλλει από το Συνταγματικό Δικαστήριο που τη θεώρησε αντισυνταγματική. Εμείς ζητούμε τροποποίηση της πράξης του 1970 που διέπει τις ευρωπαϊκές εκλογές. Εμείς ε, θέλουμε λοιπόν τροποποίηση της ε, πράξης αυτής ε, η οποία ήδη από το 1976 είχε θεωρήσει ότι θα πρέπει να γίνονται άμεσες και καθολικές εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενώ στην ε, μεγάλη πλειοψηφία τους οι ευρωπαϊκές ε, χώρες ε, οποιοδήποτε πολίτης ο οποίος έχει καταδικαστεί ενώπιον δικαστηρίου δύσκολα θα καταφέρει να βρει δουλειά στο δημόσιο τομέα ας πούμε ή ακόμα και σε αυτό το, το κοινοβούλιο, σαν ε, υπάλληλο δηλαδή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ούτε θα μπορέσει να υιοθετήσει ένα παιδί ε, ακριβώ ε, γιατί έχει ε, ποινική ε, καταδίκη, μπορεί παρόλα αυτά να εκλεγεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Να σα αναφέρω την περίπτωση του βουλευτή Μπονσινιόρε, ο οποίο ήταν και την του, του ΕΛΚ, ο οποίο έχει καταδικαστεί σε δύο χρόνια ερκτή. Ε, κάθριξη, συγγνώμη, ή επίση την υπόθεση του κυρίου Μποργέζιο, ο οποίος έχει καταδικαστεί για εμπρισμό επιβαρημένο από ρατσιστικά ε, στοιχεία. Ε, τον ε, Πατριτσέλο, ο οποίος έχει καταδικαστεί για ε, παράνομη χρηματοδότηση επίσης ε, ε, τον Ζωά Λεπέν ο οποίος έχει καταδικαστεί πολλές φορές για ρατσισμό και για παρότρινση φιλετικού μίσους. Σε αυτή την περίοδο η Επιτροπή Θεσμικών Υποθέσεων ό,τι και αν λέει ο πρόεδρος της Κάρλο Καζίνη εξετάζει μία πρόταση σε τις πράξεις του 1976 με εισηγητή τον ε, Άγγλο βουλευτή Άντριου Νταφ. Εμείς θεωρούμε ότι η τροποποίηση την οποία ζητούμε εμείς ε, μπορεί να εναρμονιστεί ε, στο πλαίσιο αυτό, όπως ακριβώς προβλέπεται και από το άρθρο 223 της συνθήκης. Δηλαδή, με τρόπο ώστε να εναρμονιστεί ο ευρωπαϊκός, η ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία παραπέμπει πάντα σε εθνική νομοθεσία αυτά τα ζητήματα με αποτέλεσμα διάφοροι καταδικασμένοι να βρίσκονται σήμερα εκλεγμένοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμεί ζητούμε απλά από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να κάνει αυτό που έχουν κάνει πάρα πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε, όπω α πούμε η Αυστρία, η Δανία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οποτεδήποτε έχει επεγγελθεί κατά δίκη υπερβαίνουσα το ένα έτο, δεν είναι δυνατόν να ε, εκλεγεί ο ενδιαφερόμενο. Χιλιάδε άνθρωποι έχουν, έχουν γράψει, έχουν στείλει επιστολέ στα μέλη τη Επιτροπή θεσμικών υποθέσεων και έχουν στείλει και την, ε, ε, ε, την αναφορά τους online σε αυτήν την Επιτροπή. Πιστεύω λοιπόν ότι κάλλιστα μπορεί να ξεκινήσει μια διαδικασία αντίστοιχη με αυτή που ξεκίνησε για τα απορρίμματα στην επαρχία της Καμπανίας. Ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να ε, δει ότι πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες και Ιταλοί πολίτες ζητούν να τροποποιηθεί ο κανονισμός που διέπει τις δυνατότητες ε, και τις προϋποθέσεις εκλογής. Ε, δεν είναι δυνατόν άνθρωποι που έχουν καταδικαστεί για σοβαρότατα αδικήματα ε, να μπορούν να, είναι, να εκλεγούν. Στις επόμενες εκλογές θα μπορούσαν ας πούμε, να φτάσουν εδώ άνθρωποι όπως ο Σαλβατόρε Κουφάνε, ο οποίος καταδικάστηκε σε δεύτερο βαθμό για επιβαρημένη διευκόλυνση συμμορίας μαφιόζης ή μαφιόζικης ή επίσης ο άλλος συνάδελφός του Μαρτσέλο Ντελούτρι, ο οποίος επίσης δευτεροβάθμια έχει καταδικαστεί ε, για ε, ε, σύσταση και συμμορία τύπου μαφίας και ο οποίος είχε αναφέρει ότι ο μαφιόζος Μαγκάνο ήταν ήρωας και των οποίων ο δικαστής ε, ε, για εγκλήματα κατά της ε, μαφίας Παύλο Μπορσελίνο είχε ορίσει ως επικεφαλής δορυφορικών οργανώσεων που βοηθούν τη μαφία στη Βόρεια Ιταλία. Θα ήθελα να κλείσω λέγοντας, αναφέροντας τα λόγια του δικαστή Μπορσελίνο, ο οποίος δολοφονήθηκε τελικά. Έλεγε λοιπόν ο Μπορσελίνο ότι και μόνο η υποψία θα έπρεπε να οδηγήσει τα κόμματα σε ένα καλύτερο ξεκαθάρισμα. Τα, τα μέλη του δεν θα πρέπει να είναι τίμια, αλλά να φαίνονται και τίμια. Και επομένω, ακόμα και αν υπάρχουν ενδείξει ανησυχητική ε, στάση, ε, πριν φτάσουμε στην πραγματική διάφραξη αδικήματο, θα πρέπει να αποκλείσουν του ανθρώπου αυτού από τα πολιτικά κόμματα. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. At the European level we have... Δύο πηγέ έχουμε. Το, εκείνη του 1986 που ορίζει τις γενικές αρχές των Ευρωπαϊκών Εκλογών και την οδηγία του 1993 που έχει σαν στόχο ότι δεν κάνει διαφορά από ποιο κράτος προέρχεται ο υποψήφιος. Όπως είπε στην πρώτη του απάντηση στον αναφέροντα κ. Κασίνη, αυτές οι δύο νομοθετικές πηγές δεν καλύπτουν τους, ε, τα προσόντα τα οποία θα πρέπει να συμμετάσχει κάποιος ή να μην συμμετάσχει κάποιος σε εκλογές. Αυτό είναι θέμα των κρατών μελών να το ορίσουν. Στην Επιτροπή Αναφορών είχαμε και στο παρελθόν αυτού του τύπου ε, αναφορές. Και στο παρελθόν καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ήταν πραγματικά αυτό το θέμα των κρατών μελών και έχει σταματήσει η κατάσταση εκεί. Θεωρώ λοιπόν ότι εάν αυτή η αναφορά γινόταν μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία των πολιτών δεν θα απαντούσα μάλλον η Κομισιόν θετικά σε αυτού του τύπου την πρωτοβουλία ε, ακόμα και αν φτάσουμε στο εκατομμύριο υπογραφές. Η κυρία Οκεν σας ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω να πω ότι το θέμα είναι πολύ δύσκολο. Γιατί αυτό που ελάχθη τώρα σχετίζεται ίσως με, αυτό, με κάτι που ελέγχθη στην ε, Δανική Βουλή. Εάν η καταδίκη είναι πάνω από ένα έτος, θα πρέπει να το τοποθετεί το Κοινοβούλιο μετά τις εκλογές για να αποφασίσει κατά πόσο αυτό το άτομο μπορεί να γίνει μέλος του Κοινοβουλίου. Εγώ είμαι πολλά χρόνια στην Δανική Βουλή και ξέρω τους κανόνες. Υπάρχει λοιπόν μια απόφαση που λαμβάνεται τότε όσον αφορά κάποιο άτομο που έχει ε, τύχη ποινική καταδίκη, χωρί να υπάρχει εκ των προτέρων ε, απαγόρευση. Είναι μια απόφαση που λαμβάνεται κατά περίπτωση από το Κοινοβούλιο. Στην Ένωση έχουμε πολύ διαφορετικέ βέβαια παραδόσει. Θα ήταν πραγματικά αδύνατο για την Δανική Βουλή να υπάρχει αυτόματη άρση ασυλίας. Ε, αν υπάρχει άρση της κοινοβουλευτικής ασύλειας, αυτό γίνεται, όπως σας είπα, κατά παρήπτωση και μέσα στα πλαίσια μιας συγκεκριμένης διαδικασίας, με νομική απόφαση. Τώρα βέβαια στην Ευρώπη δεν ξέρω είναι παντού το ίδιο. Δεν μπορεί κάποιος να προστατεύεται από την ασυλία άσχετα από το τι έχει κάνει και γιατί έχει ε, τιμωρηθεί. Οι κανόνε όμω θα διαφέρουν στην Ευρώπη και να υπάρχει μία εις βάθος απόφαση, ένας κανόνας που να ισχύει για όλους, θα οδηγήσει σε πολλά προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να το εξαιρετάσουμε. Εμένα θα μ' άρεσε ίσως να υπάρχει κάτι τέτοιο. Από την άλλη μεριά θα πρέπει να υπάρχουν κανόνες ασυλίας μεν, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω δεν μπορούμε να προχωρήσουμε πάρα πολύ. Θα πρέπει να εργαστούμε πάρα πολύ εις βάθος εκ των προτέρων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Δεν, έχουν, δεν έχω άλλους εγγεγραμμένους. Νομίζω λοιπόν ότι ακούσαμε και την ε, απάντηση για την αναφορά αυτή. Μου φαίνεται ότι η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, ήταν εξαντλητική ε, και η Σάρφα Σόουκεν η οποία μας είπε ότι είναι διαφορετική. Εδώ ασυγκρούονται διάφορες ε, δικαιοδοσίες και παραπέμπεται στο, στην ε, κατά περίπτωση ε, ανάλυση όπως υπάρχει και σε διάφορα ε, εθνικά κοινοβούλια. Αυτή η κατά περίπτωση ανάλυση γίνεται και στο, ισχύει μάλλον και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς στείλαμε και υπόμνημα στην αρμόδια καθήλυν επιτροπή, στον Προεδρό της, τον κύριο Καζίνη, Διαβιβάσαμε λοιπόν το υπόμνημα ζητώντας παρέμβαση ε, γιατί η αρχική απάντηση δεν μας είχε ικανοποιήσει. Και ο πρόεδρος Καζίνη μας απήντησε λέγοντας ότι γίνεται συζήτηση στην Επιτροπή του σχετικά με το ενδεχόμενο να ε, εκπονηθεί πρόταση τροποποιητική της πράξης του 1976 με εισηγητή όντως τον ε, Ανδρέα Νταφ ε, και για γι' αυτήν την θητεία ο ίδιος εισηγητής ο κύριος Νταφ θα εξακολουθήσει να είναι υπεύθυνο για τα θέματα αυτά. Ε, βεβαίως μπορούμε να επαναλάβουμε το αίτημά μας προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής ε, Συνταγματικών Υποθέσεων έτσι ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ε, τροποποίησης της πράξης του 1976 έτσι ώστε στις επόμενες εκλογές ενδεχομένως οι επόμενες εκλογές να γίνουν με διαφορετικό καθεστώς. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε τώρα στην αναφορά υπαριθμών 19 είναι μια αναφορά την οποία έχει υποβάλει ο πολίτης Βέρνερ Σάντιγκ είναι απόν αλλά ζήτησε να είναι παρόν στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής. Επομένως, θα δώσω αμέσως τον λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μιλήσει για την αναφορά αυτή. Ευχαριστώ. Η Επιτροπή παρακολουθεί την ε, περίπτωση, την αναφορά αυτή και διασυνοριακή αξιολόγηση για τα δύο αυτά σχέδια λαμβάνει χώρα. Το σώμα το υπεύθυνο είναι το τσεχικό Υπουργείο Περιβάλλοντος και υπάρχουν και πληροφορίες online στην ιστοσελίδα την ε, σχετική. Η αρχική διαδικασία ξεκίνησε ήδη από το 2008. Δεν έχουμε προχωρήσει πολύ, έχουμε ενημερωθεί στις 21 Ιουλίου του 2010 μόνο. Η Γερμανική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Περιβάλλοντος δεν είχε την ε, αξιολόγηση επιπτώσεων και το screening. Μέχρι τώρα το Υπουργείο έχει 11 ε, στοιχεία από κατοίκους της περιοχής και το screening θα δημοσιευθεί σε μία με δύο εβδομάδες. Ξέρουμε ότι το προκαταρκτικό screening δεν αποκλείει επιπτώσεις επί του περιβάλλοντος. Οπότε βάσει της οδηγίας Habitat θα δοθεί και η κατάλληλη συνέχεια. Τώρα, αυτός που έχει αναλάβει το έργο πρέπει να υποβάλει συστάσεις σε σχέση με την ε, έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Συνεπώς, ο χώρος αυτός θα παραμείνει σε εκκρεμότητα μέχρι να δούμε πώς θα προχωρήσει η διαδικασία και τι θα γίνει με την διαβούλευση που θα ξεκινήσει για να μπορέσει ο κόσμος να φέρει τις αντιρρήσεις του. Κύριε Ζιά, ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ την Κομισιόν για την πρώτη αυτή απάντηση. Εδώ πρόκειται για ένα πρόβλημα που έχουμε συχνά εξετάσει στην Επιτροπή Αναφορών. Δηλαδή για διαμετρολογική περιβαλλοντική περιβαλλοντικό του πρόβλημα. Θα πρέπει να δούμε τι κάνουν οι δύο αυτές χώρες και πώς θα ανταλλάσσουν τις πληροφορίες τους. Δεν υπάρχει πολλή συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Ελέγχθη ήδη ότι η, τα αυτά πάρκα θα, θα κατασκευαστούν στην τσεχική πλευρά, αλλά η περιοχή προστασίας Natura 2000 είναι από την άλλη μεριά, στη Γερμανία. Και θα πρέπει να ξέρω ότι υπάρχει και μια προϊστορία γιατί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο τα χωριά που υπήρχαν εκεί ε, καταστράφηκαν. Η φύση μας βοήθησε, μας έβγαλε δηλαδή από μια δύσκολη κατάσταση και έχουμε τώρα ένα ε, χώρο Natura 2000, μια, περιοχή προστατευόμενη περιβαλλοντολογικά. Και γι' αυτό θα πρέπει να παρακαλέσουμε η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των δύο κρατών να λειτουργήσει καλύτερα και ο αναφέρον ακριβώς στρέφεται προς εμάς με αυτή την αναφορά του και λέει ότι κοιτάξτε κάτι γίνεται στη δεχική πλευρά, δεν είμαστε πολύ ενήμεροι ούτε όσον αφορά αυτό που δημοσιεύεται, ούτε ε, αυτά που μαθαίνουμε από τον δήμαρχο της, ε, της άλλης πλευράς και όποιος γνωρίζει την ε, περιοχή αυτή και η Natura 2000 χαίρομαι που είπε η, η Κομισιόν ότι οπωσδήποτε υπάρχουν επιπτώσεις στη φύση. Τώρα θα πρέπει να δούμε μήπως θα μπορούσε τώρα ήδη να αναζηθεί μια άλλη τοποθετία Μου φαίνεται πάρα πολύ σοβαρό η αναφορά αυτή, γιατί πρέπει να δημιουργηθεί και ένα κλίμα εμπιστοσύνη. Το λαμβάνω σοβαρά υπόψη γιατί είμαι Γερμανό ε, βουλευτή, βέβαια καταρχήν, αλλά και γιατί επίση βλέπουμε πάλι μια περίπτωση όπου υπάρχουν σημαντικά προβλήματα όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος διαμεθοριακά. Και γι' αυτό το είχα ζητήσει ήδη. Θα ήθελα στην επόμενη μας συνεδρίαση να ξαναεξετάσουμε αυτή την αναφορά, παρουσία των αναφερόντων που μπορούν να μας δώσουν και πιο συγκεκριμένα στοιχεία και καλό θα ήταν και ενός εκπροσώπου της τσεχικής κυβέρνησης. Γιατί ακριβώς το κύριο πρόβλημα από πλευρά μου είναι η έλλειψη διαφάνειας. Η έλλειψη της βούλησης προς διάλογο. Ιδίως προκαταρτικά, πριν να πραγματοποιηθούν αυτές οι μεγάλες επενδύσεις και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Κομισιόν για την απάντησή της. Αλλά ακόμα υπάρχουν και άλλα πράγματα να γίνουν. Ευχαριστώ. Θα ολοκληρώσουμε την συζήτηση από αυτού του θέματος στην επόμενη συνεδρία. μας, όταν θα είναι παρόν και ο αναφέρον. Επόμενο σημείο. Έχουμε ήδη ξεκινήσει την δραστηριότητα την οποία είχαμε υποσχεθεί ότι θα αναλάβουμε. Στείλαμε επιστολή στις ελληνικές αρχές, ε, λάβαμε απάντηση η οποία θεωρώ ότι είναι εξαντλητική και απαντά στα ερωτήματα που έθεσε η αναφέρουσα. η κυρία Παλιαδέλη, ο κύριος Σαλαβράκος που παρακολούθησαν από κοντύτερα ε, το ζήτημα. Ε, συμμερίζονται οι δύο αυτοί συνάδελφοι το αίτημα να κλείσει η αναφορά αυτή γιατί πλέον και με την ανταλλαγή των τελευταίων στοιχείων δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Δεν ξέρω αν έχουμε εδώ εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο οποίος θέλει να μας πει κάτι σχετικά με το σημείο αυτό. Ο κύριος Παπούλιας. Πράγματι, εντόπισε η Επιτροπή ερευνώντας την υπόθεση αυτή και τόνισε ότι υπάρχουν ε, θέματα που θίγει η αναφέρουσα που είναι εθνική αρμοδιότητα, είναι ο αστικός σχεδιασμός, για παράδειγμα, και όσον αφορά τους ισχυρισμούς για παραβίαση περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τονίσαμε ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες αποδείξεις που να δίνει η αναφέρουσα για ε, την παραβίαση με το χτίσιμο του ξενοδοχείου αυτού στις πληροφορίες που μας έδωσε στην Επιτροπή τουλάχιστον. Δεδομένου ότι έχουμε προκαταρτικές ε, πληροφορίες από την ελληνική κυβέρνηση που δείχνουν ότι το ξενοδοχείο αυτό θα χτιστεί εν μέρη μόνο ε, στην προστατευμένη περιοχή, είναι κάτι που έχει να κάνει με την εθνική νομοθεσία. Είναι δηλαδή ε, το κράτος μέλος που πρέπει να ξεκινήσει μια περιβαλλοντική μελέτη. Συνεπώς δεν βλέπουμε εδώ παραβίαση κοινοτική νομοθεσίας. Όσον αφορά την πτυχή Natura 2000 και την παραβίαση της οδηγίας για τους οικοτόπους, και πάλι όπως σας είπα δεν έχουμε αποδείξεις από την αναφέρουσα για τις βλεβερές επιπτώσεις. Πάντω, προκειμένου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έχει την εγγύηση ότι έχει ακολουθήσει σωστά τη διαδικασία και δεδομένου ότι πρόκειται για μια περιοχή η οποία επλήγει από πυρκαγιές το 2007 και άρα είναι ευάλωτη, ζητήσαμε από τις ελληνικέ αρχές να μας δώσουν επιπλέον πληροφορίες όσον αφορά την φύση του σχεδίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Περιμένουμε λοιπόν την ενημέρωση αυτή. Αλλά από ό,τι κατάλαβα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει πληροφορίες, οπότε έτσι θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία. Μόλις έχουμε εμεί αυτές τις πληροφορίες από εσά, μας τις στείλετε, θα μπορέσουμε να κάνουμε τις δικές μας έρευνες και να κλείσουμε ενδεχομένω την υπόθεση αυτή. Θα δώσουμε λοιπόν, στη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλα τα ε, στοιχεία τα οποία έχουμε. Αυτά, δεν έχουμε τίποτα άλλο στην ημερήσια διάταξη. Ευχαριστώ ε, πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους. Θα τα πούμε στην επόμενη συνεδρίαση.